Λοιπόν, εγκρίνεται το σχέδιο μερικές διάταξης. Right. Um, as mentioned in your... Όπως αναφέρεται και στην δημοσιευθήσα ημερήσια διάταξη, το σημείο 12. Γνωμοδότηση Μαριά αναβάλλεται για τις 22 Φεβρουαρίου. Σημείο 9 η συνεδρίαση του συντονιστών ακυρούνται και η συνεδρίαση της Επιτροπής θα ξεκινήσει στις 3 το απόγευμα. Λόγω εξαιρετικών περιστάσεων, η κυρία Μπετρίς Μπεθέρα θα προεδρεύσει το απόγευμα στη συνεδρίαση. Αν δεν έχετε αντιρρήσεις, εγκρίνεται η μερίσια διατάξη. Δεν βλέπω να υπάρχουν αντιρρήσεις, θεωρείται εγκεκριμένη η μερίσια διατάξη. Σημείο 3. Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις της Προέδρου και δεν έχουμε διάφορα προς Πάμε κατευθείαν λοιπόν στην ψηφοφορία. Ανακάλυψα ότι ξέχασα την κάρτα μου ψηφοφοριών. Μπορώ διανατάσσω στις της χειρός να ψηφίσω. Είναι η πρώτη φορά, πρώτη φορά. Θα ρωτήσω εδώ να μου πούν τι θα κάνω. Με συγχωρείτε και εγώ ότι ξέχασα. Κυρία Άουκεν. Έθεσε το ερώτημα κυρία Άουκεν και δεν με ακούει τώρα να σας απαντήσω. Κυρία Άουκεν. Θέλετε να απάντηση στην ερώτησή σας. Μπορείτε. Αλλά παρακαλώ να μου ξεκαθαρίζετε πώς θα ψηφίσετε κάθε φορά. Θα έχετε πρόβλημα. Και εγώ την ξέχασα. Λοιπόν, θα είναι ηλεκτρονική ψηφοφορία. Όποιος έχει την κάρτα του, παρακαλώ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 Okay, um, quite a number of Έχουμε αρκετές συμβαστικές. Παρακαλώ λίγη ησυχία για να προχωρήσουμε. Διανατάσταση ισχυρός θα ψηφίσουμε. Για να διευκολύνουμε τους πάντες. Αν υπάρχει πρόβλημα θα γίνεται ηλεκτρονικός έλεγχος. Ωραία. Ξεκινάμε λοιπόν. σχέδιο εκθέσεως Επιτροπής Αναφόρων αφορά την ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητε του, Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή του 2014. Ψηφίζουμε τη συμβαστική τροπολογία Α. Υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική Β. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 20. Σε τρία τμήματα. 20 πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 20. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα της 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ας ελέγξουμε όμως. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική σύλλα Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 24 σε δύο τμήματα. Στην 25, 24 καταπίπτει. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Είκοσι οκτώ, τρία τμήματα. Το πρώτο τμήμα της 28 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, Αποχές. Απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα. Της 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία συμβιβαστική ε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική F ε. τενικό υπέρ κατά αποχές έλεγχος 36. Όχι. 38. Τροπολογία 38. Υπέρ παρακαλώ. Έχουμε δύο τμήματα. Τροπολογία 38. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 38.2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται και το δεύτερο τμήμα. 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Σαράντα τέσσερα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 40 συμβιβαστική G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 48 τροπολογή 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογή 49 υπέρ κατά Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 50. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία Ήτα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. σε πέντε τμήματα. Α, καταπίπτει, αλλά η 50 απορρίφθηκε. 51 λοιπόν, ψηφίζουμε την 51. Πέντε τμήματα. 51 πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έλεγχος. Θα ελέγξουμε για το τρίτο τμήμα. Το τρίτο τμήμα της 51 ελέγχουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για αυτό το κομμάτι. Απορρίπτεται. 13 με 13 ψήφους απορρίπτεται. Το, το τέταρτο τμήμα της 51 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Το πέμπτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική γιώτα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία J λατινικό υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική K υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 63 υπέρ κατά άποχες έλεγχος για την τροπολογία 63 ηλεκτρονικός έλεγχος άρχεται και πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 64 υπέρ. Σε δύο τμήματα. 64 πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 64 δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη. Τροπολογία 1. Της αιτιολογικής σκέψης C. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Θα κάνουμε έναν έλεγχο. Για την αιτιολογική σκέψη C. Τροπολογία 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία L, λατινικό υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Πέντε. Για την τελική σκέψη L, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τοπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τοπολογία 10 υπέρ κατά άποχες έλεγχος λοιπόν άρχεται και πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται έντεκα σε δύο τμήματα έντεκα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά σας παρακαλώ άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται Έχουμε και άλλες δύο ψηφοφορίες. The next vote is the, on the Η επόμενη ψηφοφορία αφορά την κύρωση της συνθήκης του Μαρακές με βάση τις αναφορές που ελήφθησαν. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Η επόμενη ψηφοφορία που έχουμε αφορά τι κατευθυντήριε γραμμέ τη Επιτροπή Αναφορών. Ηλεκτρονική ψηφοφορία, παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα. Ωραία, εγκρίνεται. Ευχαριστώ κύριε και κύριοι για την υπομονή σα. Right. Um, we will be... Ωραία, λοιπόν, θα ξεκινήσουμε αμέσω το εργαστήριο. Καλώς ορίζω τον πρόεδρο του εργαστηρίου, την κυρία Καπεσόν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 morning, buenos días. Bueno, pues, si os parece... Λοιπόν, αν ε, συμφωνείτε, ξεκινούμε το... το Έχουμε μόνο μέχρι το 12.30. Ξεκινάμε λοιπόν ε, αυτή τη συνεδρία εργασία, workshop. Πρέπει λοιπόν να έχουμε επαρκή χρόνο για να ακούσουμε τους εμπειρογνώμονες μας και να ακούσουμε. Καταρχά θέλω να ευχαριστήσω του για την παρουσία τους που ήρθαν εδώ να μας ενημερώσουν για ένα θέμα που ανησυχεί το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι θα δώσουν την άποψή τους, τη διαφορετική τους απόχρωση, αλλά είναι ένα θέμα που μας απασχολεί όλους εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μας ενδιαφέρει πολύ να ακούσουμε την άποψή σας ως εμπειρογνώμονες, ως επαγγελματίες του κλάδου, οπωσδήποτε θα διευκρινίσει το σημαντικό αυτό ζήτημα. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας, σας ευχαριστώ για την καλοσύνη σας που δεχτήκατε την πρότασή μας, που δεχτήκατε να έρθετε χωρίς καμία αμοιβή. Σας ευχαριστώ πολύ και η παρουσία των συναδέλφων και πολλών άλλων ε, παρευρισκομένων δείχνει πόσο ενδιαφέρον υπάρχει για το θέμα αυτό. Δεν θέλω να πω περισσότερα διότι η Επιτροπή Αναφορών όπως ξέρετε λαμβάνει πολλές αναφορές ε, κάθε χρόνο γύρω στις 3.000 αναφορές λαμβάνουμε προσπαθούμε να δώσουμε απαντήσεις προσπαθούμε να τις ε, συνοψίσουμε σε συγκεκριμένες κατηγορίες και γι' αυτό κάνουμε ε, μια προσπάθεια για να ενημερωθούμε ε, είτε μέσω ακροάσεων είτε μέσω αποστολών. Το θέμα της υγείας οπωσδήποτε απασχολεί πολλές ε, αναφορές και κυρίως αναφέρονται αυτές οι αναφορές στα προβλήματα πρόσβασης στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ιδίως στα καινούργια προϊόντα. Τέτοιου τύπου αναφορές λαμβάνουμε εδώ σε Επιτροπή Αναφορών. Η συζήτηση για την βιωσιμότητα του συστήματος ε, υγείας ε, απασχολεί όλα τα κράτη-μέλη και έχει αποκτήσει πολύ περισσότερη σημασία λόγω της συγκυρίας οικονομικής κρίσης. Έχουν γίνει περικοπές στον τομέα της υγείας σε πολλές χώρες και κυρίως βέβαια σε εκείνες που υπέστησαν ε, περισσότερο την οικονομική κρίση. Αυτό το θέμα θα μας απασχολήσει εάν μπορούμε να εγγυηθούμε με τους προϋπολογισμούς και τις περικοπές που έχουμε την βιωσιμότητα του συστήματος αυτού γιατί υφίσταται και νέες προκλήσεις το σύστημα υγείας όπως για παράδειγμα οι νέες τεχνολογίες. Θέλουμε λοιπόν την άποψη των εμπειρογνωμών. Βεβαίως ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, τα άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεν έχουν πλήρες αρμοδιότητες για το θέμα αυτό, αλλά παρόλα αυτά θέλουμε να συζητήσουμε το θέμα αυτό γιατί θεωρούμε ότι έχουν ρόλο να παίξουν και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί γιατί η σύμβαση της ε, συνθήκη της Λισαβόνας συγγνώμη, αναφέρεται στα θεμελιώδη δικαιώματα υπάρχει και ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης που έχει επικυρωθεί από την συντριπτική πλειοψηφία των κρατών μελών και αναφέρεται στο δικαίωμα προστασίας της υγείας και λέγεται ακριβώς σε αυτόν τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη ότι πρέπει να εγγυηθούμε την πρόσβαση στην ε, υγεία και την περίθαλψη σε όλους τους κατοίκους των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει λοιπόν επαρκής βάση για να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό και υπάρχει και μία άλλη βάση. Νομίζω ότι οι πολίτες μας στο σύνολό τους θεωρούν ότι το κοινωνικό κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάτι το οποίο θεωρούν αναφέρετο δικαίωμα. Και φυσικά το δικαίωμα στην υγεία είναι αναφέρετο τμήμα της κοινωνίας αυτής και της ε, προστασίας των ε, βασικών δικαιωμάτων. Άρα είναι αναγκαίο και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να απαντήσουν στις ερωτήσεις που τους τίθενται. Δεν θέλω φυσικά εγώ να σας απασχολήσω περισσότερο, αλλά θέλω να τονίσω ότι και εγώ ενδιαφέρομαι πάρα πολύ για να ακούσω τους ε, ομιλητές μας. Πρώτα απ' όλα, θα έχουμε δύο τμήματα λοιπόν. Το πρώτο τμήμα θα ασχοληθούμε με το δικαίωμα ε, στην υγεία και πώς έχουμε φτάσει στη σημερινή κατάσταση των συστημάτων περίθαλψης και πώς θα ε, μπορέσουμε να βελτιώσουμε την ε, προστασία της υγείας. Έχουμε λοιπόν εδώ τον κύριο, κύριο Στρέκερ, ο οποίος είναι καθηγητής ε, για θέματα υγείας του Πανεπιστημίου του Ντάραμ, που θα μας μιλήσει για τη σημασία των πολιτικών επιλογών στα θέματα υγείας. Και του δίνω απευθείας τον λόγο. Δυστυχώς ο καθηγητής είναι εκτός μικροφώνου, και τον ακούμε καλά. Good. Καλώς είναι τιμή μου να παρίσταμαι. Σε μεγάλο ποσοστό είμαι εδώ λόγω ενός βιβλίου που ένα συνάδελφος και εγώ δημοσίευσαμε πέρσι. Πώς οι πολιτικές μας αρρωσταίνουν. Υπότιτλος είναι οι ε, διάφορες επιδημίες θα εστιαστώ όχι μόνο στα συστήματα τα υγειονομικά, όσο στους τρόπους με τους οποίους το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον έχει αυξήσει την ανάγκη για τα συστήματα περίθαλψης. Θα ρίξω μια ματιά στην ύφεση σε σχέση με την σημότητα. Υπάρχει νέα συνένεση όσον αφορά το θέμα αυτό, ότι η ανεργία και η ύφεση τελικά βελτιώνουν τα αποτέλεσμα σε αφορά την υγεία βραχυπρόθεσμα. πρόθεσμα διότι πίνουν λιγότερο και καπνίζουν λιγότερο οι άνθρωποι και οδηγούν και λιγότερο. ταυτόχρονα όμως οδηγούμεθα και σε μια αύξηση από ό,τι βλέπουμε στην ευρωπαϊκή εμπειρία, οδηγούμεθα σε αύξηση πολύ μεγάλη στις αυτοκτονίες, στον αριθμό αυτοκτονιών. Και αυτό ταιριάζει με πρώτερα αποτελέσματα. Αλλά είναι πιο τονισμένα τα αποτελέσματα τώρα. Να δείτε τώρα τις τάσεις, τη αυτοκτονία στην Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση τον 12 και τον 15 πριν και μετά την οικονομική κρίση. Τιμές 2007 η τιμή είναι ένα, Βλέπετε το, το γράφημα. Αυτοκτονίες και ανέργεια, ανεργία στην Ελλάδα πιο συγκεκριμένα. Ένα δραματικό παράδειγμα στο οποίο θα επιστρέψω λίγο αργότερα. Και εδώ έχουμε αυτοκτονία και ε, ανεργία στην Αγγλία. Βλέπετε δραματικά σχήματα στα γραφήματα αυτό δεν σημαίνει ότι οι θέσεις σου κάνουν καλό στην υγεία. Ε, υπάρχουν θετικές και αρνητικές συνέπειες και οι μεν μπορεί να ακυρώνουν τις δε και να καλύπτουν τις αρνητικές συνέπειες κυρίως σε ευάλωτα τμήματα του πληθυσμού όπως σε άτομα υψηλού κινδύνου όσον αφορά την ε, ανεργία. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Άλλο παράδειγμα προέρχεται από την πρόσφατη μελέτη που, συνεργο... που και αν κοστείτε βραβείο Νόμπελ είχε συγγράψει μαζί με μένα. Στο αριστερό τμήμα του γραφήματος βλέπετε τι τάσει στη θνησιμότητα εν γέννη από όλα τα αίτια σε ηλικιακή ομάδα ε, με σύλλικες και συγκρίνουμε διάφορες χώρες και είναι στον πληθυσμό των λευκών στις ΗΠΑ σε σύγκριση με τους λευκούς στην ΗΠΑ. Ξεκινάμε το 2000 πριν την κρίση και βλέπουμε ότι έχουμε δραστική αλλαγή όσον αφορά τη θνησιμότητα στην ομάδα αυτή και βλέπουμε την θνησιμότητα από ασθένειες και από απελπισία δεξιά στο δεξί γράφημα για αρκετές ηλικιακές ομάδες. Στους ε, λευκούς μη ισπανικής καταγωγής, ισπανόφωνης καταγωγής, μπορούμε να πούμε ότι αυτή η ομάδα πιθανότατα να πλήττεται όλος ιδιαίτερος από την ανεργία, οικονομική ανασφάλεια και φαίνεται σαν την αρχή μιας κρίσεως ε, τύπου ρωσικού όσον αφορά την σημότητα. Λοιπόν, ποιοι είναι οι όροι και περιορισμοί. Άλλη προπτική βραχυπρόθεσμη, άλλη μακροπρόθεσμη, βλέποντας τι συνέπεια έχει η αύξηση της μακροπρόθεσμης ανεργία. Ένα άλλο θέμα είναι ότι η θνησιμότητα είναι, δύσκο είναι εύκολο να προσμετεθεί σαν δείκτης. Ε, μπορεί να πει κανείς ότι πέθανε, είναι εύκολο να διαπιστώσει ότι πέθανε, αλλά είναι πολύ ε, θα έλεγα, δεν δείχνει λεπτομέρειες πώς επηρεάζεται η υγεία των παιδιών στην ύφεση που δεν θα φαίνεται τόσο πολύ στα στοιχεία θνησιμότητας παρά μόνο μετά την πάροδο δεκαετιών. Άλλη μια διάσταση του προβλήματος αφορά την ύφεση και τις ανισότητες στον τομέα της υγείας. Ίσως τα αποτελέσματα στην υγεία επηρεάζονται από εθνικές πολιτικές που ποικίλουν και εδώ ερχόμαστε άμεσα στο θέμα του σημερινού εργαστηρίου μας. Ε, γνωρίζουμε ότι υπήρξαν κάποιες αλλαγές και βραχυπρόθεσμα και εξαρτώνται από τον τρόπο με τον οποίο οι χώρες αντιδρούσαν στην οικονομική κρίση και γνωρίζουμε από την μακροπρόθεσμη έρευνα ότι οι πολιτικές του κράτους προνοίας έχουν προστατευτικό αποτέλεσμα και το προστατευτικό αποτέλεσμα ποικίλει ανάλογα με την πολιτική. Πού το πάμε με όλα αυτά τα στοιχεία. Λοιπόν, βλέπουμε ένα πρόσφατο άρθρο και οι παραπομπές βρίσκονται στη διαφάνεια και βλέπετε ε, το πλαίσιο στο οποίο εξετάζουμε τη συνέπειση την υγεία που έχει η οικονομική κρίση και τι βλέπουμε ότι σε κάθε επίπεδο, σε κάθε στάδιο η έκθεση, η διαδικασία και τα αποτελέσματα. Πολιτικοί παράγοντες, πολιτικές επιλογές έχουν σημασία. Τα συστήματα προνοίας ε, είναι μία από τις επιρροές, πολύ σημαντικός παράγον, όμως. Ε. Ποιο είναι το βασικό μήνυμα. Ότι οι επιλογές όσον αφορά την πολιτική που ακολουθείτε είναι πολύ σημαντικές και ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης μπορεί να μετριαστεί από την κοινωνική πολιτική ή να επιδεινωθεί από τη λιτότητα και περικοπές όσον αφορά την πρόνοια. Διάφοροι συνάδελφοι έδειξαν ότι υπάρχει στατιστικός συσχετισμός μεταξύ των ποσών που δαπανούν οι χώρες για τα προγράμματα της ενεργού αγοράς εργασίας και των ποσοστών αυτοκτονίας. Και το βασικό μήνυμα που σας δίνω είναι ότι η δημόσια χρηματοδότηση αφορά τη δημόσια υγεία άμεσα. Ε, και απόδειξη αυτού του σημείου απορρέει από μια μελέτη που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Η μελέτη αυτή εξέτασε ξεχωριστά τις συνέπειες που έχει η ύφεση και τα προγράμματα λιτότητας πώς επηρεάζουν διάφορα ποσοστά ε, Σε 23 ευρωπαϊκές χώρες βλέπουμε θνησιμότητα που είναι ένας πολύ γενικός δείκτης mm. και ε, βλέπετε εδώ τα πορίσματα που σας προανέφερα, που δείχνουν τα πορίσματα. Το εξής, όταν εξετάζουν ενεργή αυτή καθεαυτή απομονωμένη, τίνει να έχει κάποια μείωση. Να, βλέπετε, να μειώνει τη θυσιμότητα Βλέπετε τη μειωμένη θυσιμότητα στο αριστερό τμήμα του γραφήματος. Αν δείτε τις συνέπειες της λιτότητας που προσπαθεί να διορθώσει και κάνοντας τη διόρθωση την ανεργία. Η ανεργία θεωρείται σαν μια σταθερά και βλέπετε μια πολύ σημαντική αύξηση στη θνησιμότητα στο δεξί κομμάτι. Δυστυχώς το επιστημονικό έγγραφο που εξηγεί την πλήρη μεθοδολογία δεν έχει ακόμα δημοσιευτεί, αλλά άλλες στοιχές της μελέτης έχουν δημοσιευτεί. Και έγιναν αποδεκτές από την εξέταση των ομοτήμων. Τώρα κάποιες συγκεκριμένες μελέτες συγκεκριμένες χώρες. Πρώτη, πιθανότατα γνωστή περίπτωση είναι η Ελλάδα στην Ελλάδα η επέτηση για ένα νοτατόριο όσον αφορά τις δημόσια δαπάνες για την υγεία ήταν ένα κομμάτι ε, του, του, της, ε, του μνημονίου. Ε, λοιπόν, το status quo δεν ήταν δυνατό να παραμείνει, αλλά οικονομολό, ο Τζόζεφ Στίγκλετ μεταξύ μου άλλων είχε πει γιατί θα πρέπει να πληρώνουν οι πολίτες για προγράμματα που κυρίως ε, ευνοούν τους πιστωτές του δημόσιου τομέα. Αυτό είναι ένα σαφές παράδειγμα ενός συστήματος υγείας το οποίο επιδεινούται και σχετίζεται αυτή η επιδείνωση άμεσα με τη λιτότητα. Και η μείωση του, της περίθαλψης για την ψυχική υγεία είναι κάτι που δεν θες να κάνεις όταν η κατάσταση όλη ευνοεί την αύξηση των αυτοκτονιών. Και έχουν γραφεί διάφορα άρθρα πάνω στο θέμα και προειδοποιούν για τις συνέπειες που έχουν αυτά τα μέτρα. Άλλη μελέτη συγκεκριμένη, Ισπανία και Πορτογαλία, έχουμε διάφορα αποτελέσματα όσον αφορά τις αλλαγές συστηματαγίας. Χρειάζονται τα αποτελέσματα και ο αντίκτυπος ε, σε διάφορους δείκτες κάποιο χρόνο για να φανούν. Αλλά ένα έγγραφο δημοσιεύτηκε μόνο στο, στη Διεθνή Εφημερίδα των Υγειονομικών Υπηρεσιών ε, δείχνει ότι υπάρχουν αρνητικά αποτελέσματα μεταξύ των ευάλωτων τμήματων του πληθυσμού αυτών των, πλη... των τμήματων πληθυσμού που ανέφερα, όπου τα αποτελέσματα να μην φαίνονται σε θνησιμότητα, αλλά σε άλλες μεταβλητές. Αυτό ίσως να είναι κάπως να μην είναι τόσο γνωστό, αλλά είναι από εκεί που μένω, στη χώρα στην οποία μένω και δουλεύω, στο Ηνωμένο Βασίλειο, που η κυβέρνηση προτείνει να μειώσει τη δημόσιες δαπάνε σαν ποσοστό του ΑΕΠ στα επίπεδα της δεκαετίας του 30 πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πριν δημιουργηθεί το Εθνικό Σύστημα υγεία. και, και έχει, έχει μικρύνει το κόστος σε επίπεδα που υπήρχαν πολύ πριν, πριν πολλές γενιές και επηρεάζει πολλές περιοχές και πολλά τμήματα του πληθυσμού αυτή η μεγάλη περικοπή. Εδώ βλέπετε ένα γράφημα που στον κάθε τάξονα έχουμε το, το ποσό ε, που θα αφαιρεθεί για κάθε ενήλικα εργαζόμενο ε, στην, στον Ηνωμένο Βασίλειο και στον οριζόντιο άξονα βλέπουμε τη στέρηση. Οι πιο στερημένες περιοχές, οι πιο φτωχές περιοχές είναι στο άκρο δεξιό του Ηνωμένου Βασιλείου και βλέπετε μία τάση τα αποτελέσματα πλήττουν τους φτωχότερου ανθρώπους και τις φτωχότερε περιοχές πιο σκληρά. Εδώ η λιτότητα δεν πλήττει μόνο τους πιο φτωχούς ανθρώπους και τις περιοχές, αλλά πλήττει και τους, τις πιο ασθενείς περιοχές, τις νοσούσες περιοχές. Στο γράφημα αυτό, στον κάθετο άξονα, βλέπετε την, την τιμή των περικοπών προς την τοπική αυτοδίκηση κατά κεφαλή, κατά κάτοικο δηλαδή, και οριζόντια πρώιμη θνησιμότητα, κατά 100, ανά 100.000 του πληθυσμού. Και οι, πιο, οι, νοσούσες περιοχές, οι πλέον νοσούσες περιοχές είναι προς τα δεξιά και βλέπετε ότι υπάρχει ένας σαφής ε, συσχετισμός στα στοιχεία. Λοιπόν, τα μαθήματα και τα συμπεράσματα, η οικονομική ανισότητα και η κοινωνική πολιτική ε, επηρεάζουν την κατάσταση, το ξέρουμε από τις μελέτες και το, τις του Κρίγκερ και άλλων στις Ηνωμένες Πολιτείες και διάφορα αποτελέσματα στον Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, κάπως εδώ πιο χαλαρά ερμηνεύσαμε τα στοιχεία σε αυτό το γράφημα, διότι από επιλεγήσεις περιόδους πήραμε τα στοιχεία και όλα τα στοιχεία δεν έχουν την ίδια διάρκεια και δεν έχουμε την ίδια ποιότητα στα στοιχεία, αλλά βλέπετε ότι υπάρχει σαφή στάση κυρίως στο μεταγενέστερο κομμάτι ε, ότι οι ανισότητες αυξάνονται προς το τέλος της δεκαετίας του 70 και αυτό που είναι ενδιαφέρον από αυτή τη γραφική παράσταση είναι όταν το συγκρίνεις με, μια, με ένα γράφημα που δείχνει τάσεις σε οικονομικές ανισότητες ξεκινώντας ξανά περίπου τα τέλη της δεκαετίας του 70 και βλέπεις ε, τους συσχετισμούς ε, που είναι αρκετά παρεμφερείς. Για να επαναλάβω λοιπόν αυτό που έλεγα, τα δημοσιονομικά, δημόσιες δαπάνες ε, επηρεάζουν άμεσα τη δημόσια υγεία, η λιτότητα κατ' παρελθόν και τώρα είχε αποδεικνυόμενα αρνητικά αποτελέσματα για την υγεία. Και ο Ντέφιγκ Στόγκλερ και άλλοι ανέφεραν αυτό που συζητούμε σήμερα. Δηλαδή ότι τα αποτελ... είναι ένα πείραμα ε, μεγάλης κλίμακας σε ανθρώπους, ανθρώπινο πληθυσμό που δεν έχει συμφωνήσει να διεξαχθεί το, το πείραμα. Λοιπόν, ζητώ συγγνώμη αν πήρα κάποιο χρόνο τον άλλο μιλητή ή κάλυψα κάποια στοιχεία του επόμενου μιλητή. Δεν συγκρίναμε τι σημειώσει μα προηγουμένω. Θα έλεγα ότι η λιτότητα υπονομεύει το δικαίωμα στην υγεία στην Ευρώπη, κυρίω διότι αντιβαίνει ε, της, ε, την αρχή της μη παναχώρησης όσον αφορά τα κεκτημένα της υγεία. Ο Κλέρ Μπράμπρα, η Κλέρ Μπράμπρα και εγώ ε, έχουμε και άλλου υποστηριχτές. Το 2013 ε, είπα το εκπρόσωπο τα ανθρώπινα δικαιώματα το ΙΕ είπε τα ίδια πράγματα λίγο πολύ, Διέταξα πάρα πολύ υλικό τάχιστα για να παραμείνω εντός των χρονικών ε, περιθωρίων, αλλά προσβλέπω στις ερωτήσεις σας και θα δώσω το λόγο στον επόμενο παρουσιαστή, στον επόμενο μιλητή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Στράκερ. Πολύ ενδιαφέρουσα η ομιλία σας, ιδίως αυτό που είπατε για τις επιπτώσεις μέσω και μακροπρόθεσμα των περικοπών που διαπιστώνουμε στις χώρες ε, στις οποίες αναφερθήκατε και εσείς, οι Ηνωμένες Πολιτείες ε, και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η κυρία Λίλιαν Κέλλη τώρα που είναι ε, εμπειρογνώμων για τέτοια θέματα που θα μας μιλήσει για τις επιπτώσεις της κρίσης ε, στο δικαίωμα πρόσβαση στην υγεία σε διάφορες χώρες της Ένωσης, παρελθόν, παρόν και ε, προοπτικές για το μέλλον. Καλημέρα σας. Έχω έρθει από την Ηλιό για να σας προσθέσω μια μελέτη που κάναμε πέρυσι για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τις επιπτώσεις της κρίσης για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Εγώ θα παρουσιάσω τη μελέτη όσον αφορά τις επιπτώσεις της κρίσης στην πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη. Ε, εξετάζουμε επιλεγμένα, θεμελιώδη δικαιώματα σε επιλεγμένα κράτη-μέλη, προσέχοντας ιδιαίτερα τη φύση και τις επιπτώσεις των μέτρων που έλαβαν τα κράτη-μέλη μόλις ξεκίνησε η οικονομική κρίση να σας παρουσιάσω τη μέθοδο που χρησιμοποιήσαμε για τη μελέτη μας επειδή η κρίση δεν έπληξε ε, με την ίδια ένταση όλα τα κράτη-μέλη εξετάσαμε την κατάσταση σε 7 κράτη-μέλη που επλέξαν ιδιαίτερα από την ε, οικονομική κρίση. Τα κράτη αυτά δίνουν μια αντιπροσωπευτική εικόνα όλης της κατάστασης ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και περιλαμβάνοντας αυτά κράτη-μέλη που έλαβαν χρηματοοικονομική στήριξη και άλλα που όχι και με διαφορετικά ε, συστήματα. Τα δικαιώματα που επλήγησαν περισσότερο κατά την οικονομική κρίση ήταν τα οικονομικά και ε, κοινωνικά δικαιώματα και αυτά που επλήγησαν περισσότερο βάσει ε, τα εξετάσαμε σε όλα τα κράτη-μέλη και το δικαίωμα για την υγειονομική περίθαλψη ήταν ένα από αυτά που πλήξαν περισσότερο. Όπως βλέπετε τα κρατημέλη που επιλέξαμε ήταν το Βέλγιο, η Κύπρος, η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Ισπανία. Και τα δικαιώματα που επιλέξαμε σε αυτά τα κρατημέλη ήταν το δικαίωμα ε, για την εκπαίδευση, για υγειονομική περίθαλψη, για εργασία, για συνταξιοδότηση, για πρόσβαση στη δικαιοσύνη και η ελευθερία έκφρασης και η ελευθερία του συνεταιρίζεστε. Του συνερχίστε, συγγνώμη. Όπω βλέπετε λοιπόν το δικαίωμα για υγειονομική περιθάλψη ήταν από αυτά που επλήξαν περισσότερο κατά την οικονομική κρίση. Η κρίση και τα μέτρα λιτότητα επηρέασαν και άλλα ε, δικαιώματα στα κράτη-μέλη. Εδώ θα δούμε μια επισκόψη των δικαιωμάτων που επηρεασαν συγκεκριμενα συγκεκριμένα, ε, συγκεκριμένα κράτη-μέλη, για παράδειγμα το δικαίωμα στην πρόσβαση σε νερό, το δικαίωμα εργασία και ελευθερία ενημέρωση. Δεδομένη τη συνεχώ μεταβαλλόμενη κατάσταση στα κράτη-μέλη, κατέστη απαραίτητο να καθορίσουμε μια ημερομηνία διακοπή ε, για ε, την ανάλυση και τι εκθέσει που παρουσιάσαμε και στι ε, εκθέσει των 7 χωρών. Αποφασίσαμε λοιπόν ότι αυτή η ημερομηνία θα ήταν η 30 η Ιουνίου του 2014. Και σε περίπτωση που κάτι σημαντικό συνέβαινε μετά από αυτή την ημερομηνία μέχρι την οριστικοποίηση τη μελέτη το Φεβρουάριο του 2015 θα είχαν συμπεριληφθεί. Οι μεθόδοι έρευνας που χρησιμοποίησαν βασίστηκαν στους διαθέσιμες πηγές ε, βάσει βιβλιογραφίας ε, και επίσης είχαμε και διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Τώρα, όσον αφορά το δικαίωμα για πρόσβαση στην υγειονομική περίθαψη, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Διεθνού Συμφώνου για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα, ε, αναφέρεται ότι το δικαίωμα καθενός ε, στο υψηλότερο πιθανό επίπεδο ε, σωματικής και πνευματικής υγείας πρέπει να διασφαλίζεται. Η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών αναφέρει ότι το δικαίωμα για την υγειονομική περίθαλψη πρέπει να, είναι, ε, να χαρακτηρίζεται από διαθεσιμότητα, προσβασιμότητα, αποδεκτό και ποιότητα. Ακόμη και πριν την κρίση είχαν αλλάξει οι υποδομές στον τομέα της υγείας με το ξέσπασμα της κρίσης οι μεταρρυθμίσεις του τομέα έγιναν πιο επίγουσες Είχε υπάρξει υπόσχεση ότι θα ήταν φθηνότερες υπηρεσίες και καλύτερες, αλλά η κρίση θεωρήθηκε δηλαδή ως ευκαιρία για να γίνουν κάποιες μεταρρυθμίσεις που έπρεπε να είχαν γίνει πριν καιρό. Σε όλα τα κράτη-μέλη που εξετάσαμε εισήχθησαν ε, μέτρα όσον αφορά την πρόσβαση ε, ανάλογα με τις συνθήκες λιτότητας και της οικονομικής κρίσης ενώ δεν γνωρίζουμε στο Βέλγιο να υπήρξαν απτά μέτρα πάγωσε ο υπολογισμός της ε, υγειονομικής περιθέλψης ε, αλλά εισήχθησαν μέτρα βελτίωσης της πρόσβασης. Για παράδειγμα υπήρξε ένα τέλος απαγόρευση, ένα ε, τέλος για νοσοκομιακή περιθέλψη και διπλά δωμάτια. Σε κάποια άλλα κράτη-μέλη έγιναν σοβαρές περικοπές στι σχετικές δαπάνες. Για να δούμε τα μέτρα λιτότητα που εφαρμόστηκαν στα κράτη-μέλη, μεταξύ αυτών βλέπουμε μεταρρυθμίσεις στο υγειονομικά συστήματα, περιορισμένη πρόσβαση στην υγειονομική περιθάλψη, για παράδειγμα στην Ισπανία η πρόσβαση στην υγειονομική περιθάλψη από εντελώ δωρεάν μετατράπηκε σε ένα σύστημα που βασιζόταν ε, στην κατάσταση απασχόληση του εν λόγω ατόμου. Τα τέλη συμμετοχή επίση εισήχθησαν για ορισμένε υπηρεσίε, για παράδειγμα για την πρωτεύουσα βοήθεια, για κάποια τεστ, για κάποιε επίγουσε επισκέψει και επίση ε, αυξήθηκαν και οι συμμετοχέ. Αναδιοργανώθηκαν τα νοσοκομεία και οι προμηθευτέ υπηρεσιών υγεία ε, έγιναν παρεμβάσεις στο κόστος των φαρμάκων και λοιπόν υπηρεσιών και κάποια από αυτά τα μέτρα βασίστηκαν σε παρεμβάσεις ε, για παράδειγμα στην τιμή των γενώσιμων φαρμακών από τα κράτη-μέλη ε, τα οποία όρισαν μέγιστες τιμές πολύ στα φαρμακεία επίσης και άλλα μέτρα ήσυξαν. για παράδειγμα στην Πορτογαλία έγιναν περικοπές στη φοροαπαλλαγή για την υγειονομική περίθαλψη ενώ στην Ιρλανδία αυξήθηκε η ιδιωτική ε, ασφαλιστική κάλυψη. Όλα αυτά τα μέτρα λιτότητας επηρέασαν ε, χαρακτηριστικά τα δικαιώματα στην υγειονομική περίθαλψη στα κράτη-μέλη. Οι περικοπές ε, των δαπανών στον τομέα παρεμπόδισαν ορισμένες ομάδες από τον έχουν πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη. Κάποια μέτρα επέβαλαν περισσότερο οικονομικό φόρτο σε κάποιους πολίτες. Για παράδειγμα, ε, τα τέλη επίσκεψης αυξήθηκαν και επίσης αυξήθηκε και το κόστος των υπηρεσιών υγείας. Μειώθηκε επίσης ο αριθμός του προσωπικού και των ε, υποδομών που υπήρχαν διαθέσιμα. Επίσης ε, ένα εμπόδιο παρατηρήθηκε στην πρόσβαση, μειώθηκε ο αριθμός των κρεβατιών στα νοσοκομεία, σε ορισμένα κράτη-μέλη, αυξήθηκαν οι χρόνοι αναμονής για ραντεβού, ιατρικές εξετάσεις και χειρουργία. Επίσης, λόγω του επιπλέον οικονομικού φόρτου και των ε, μεγαλύτερων ε, ληστών αναμονής, ε, κάποιοι αναζήτησαν εναλλακτικές, χρησιμοποιώντας ιδιωτική υγειονομική παράθλιψη ή απευθυνόμενοι σε μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Δηλαδή στην Ελλάδα, για παράδειγμα, πολλοί κόσμοι πήγε σε κοινωνικέ κλινικέ, κοινωνικά φαρμακεία που στελεχώνονται από εθελοντές. πολλοί κόσμος επειδή δεν μπορούσε να πληρώσει ε, το τέλος των φαρμάκων ή της ιατρικής περιθέλψης ε, ή επειδή ήταν πολύ μακριά οι τόποι περιθέλψης ε, αντιμετώπισαν προβλήματα. Λόγω των περικοπών επηρεάστηκαν και τα προληπτικά μέτρα και τα μέτρα προστασίας. Για παράδειγμα, μειώθηκε ο αριθμός παιδιών που εμβολιάζονταν. Επίσης έγιναν παρεμβάσεις στην αγορά των φαρμάκων λόγω λήψεων και προμήθειας ορισμένων φαρμάκων. Όλα αυτά τα μέτρα λιτότητας επηρέασαν πολύ άσχημα ευάλωτες ε, ομάδες του πληθυσμού. Για παράδειγμα τους φτωχούς, τους ε, αστέγους, τους ε, ηλικιωμένους, ανθρώπους με αναπηρίες και τους συγγενείς τους και τις γυναίκες. Όλοι αυτοί επηρεάστηκαν πολύ αρνητικά από τα μέτρα που επιβλήθηκαν. Να περάσω τώρα σε μια μελέτη περίπτωση τη Ιρλανδίας, επειδή εγώ υπήρξα συντακτηρέα τη Ιρλανδική Έκθεση για τις επιπτώσει τη κρίση στα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ιρλανδία ω αποτέλεσμα τη οικονομική κρίση, Τα μέτρα λιτότητας που εφαρμόστηκαν επηρέασαν σημαντικά το δικαίωμα πρόσβαση στην οικονομική περίθαλψη. Πολλοί πολίτε πιστεύουν ότι αυτό είναι ο τομέα όπου οι περικοπέ έχουν τα χειρότερα αποτελέσματα. Τα μέτρα λιτότητα που εφαρμόστηκαν συμπεριλάμβαναν περικοπές χρηματοδότησης στην δημόσια χρηματοδοτούμενη υπηρεσία υγείας της Ιρλανδίας, επίσης ε, μείωση ε, των ε, προσλήψεων στον τομέα αυτό, περικοπές προσωπικού, αυξημένα τέλη επίσης επιβλήθηκαν σε ασθενείς για κρεβάτια, για περίπτωση ατυχημάτων ή επιγόντων περιστατικών, ε, για ε, ιατρικές συνταγές ε, και τα λοιπά. Επίσης αυξήθηκε το κόστος της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας. Πολύ σημαντικό ζήτημα αυτό. Διότι πολλοί κόσμοι βασίζεται στην ιδιωτική ασφάλεια στην Ιρλανδία. Και επίσης μειώθηκαν επίσης οι δαπάνες για την ε, ψυχική υγεία. Όλα σε αυτές τις περικοπές επηρέασαν σημαντικά την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη. Το σχέδιο εξυπηρέτησης του 2015 προέβλεπε ε, το κλείσιμο από 555 έως 898 κρεβατιών σε γεροκομεία λόγω περικοπών οι γενικά παρεχόμενες δωρεάν υπηρεσίες όπως επισκέψεις ε, νοσοκόμων σε νεογέννητα, εμβολιασμοί ε, περιορίστηκαν σημαντικά. Οι λίστες αναμονής επίσης να αυξάνονται γεωμετρικά και όλα αυτά σχετίζονταν με τις περικοπές της χρηματοδότηση ε, τις περικοπές χρηματοδότησης και επίσης ε, υπήρξαν και περικοπές ε, με αποτέλεσμα προβλήματα στην κατοίκον περίθαλψη και σε όλη την αγορά της υγειονομικής περίθαλψης. Πάνω από 200.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν την ιδιωτική ε, ασφάλιση υγειονομικής περίθαλψης από το 2008 και επίσης επιβλήθηκαν επιπλέον δαπάνες. Για παράδειγμα το 2013 κάθε άτομο πλήρωνε, κατέβαλε περίπου 100 ευρώ σε επιπλέον δαπάνες για την πρόσβαση σε περίθαλψη και ε, ε, συνταγογραφούμενα φάρμακα. Τέλος, θα ήθελα να προτείνω κάποιες συστάσεις που αναδείχθηκαν ε, εντός μελέτης και που θα έπρεπε να επιβληθούν ανεξάρτητα του εύρους του σκοπού οποιοδήποτε μέτρο που εφαρμόζεται η γνωμική περίθαλψη πρέπει ανά πάσα στιγμή να συμμορφώνεται με τα πετούμενα πρότυπα διαθεσιμότητας ε, της ε ε, ε, ε, φθηνής τιμής και ποιότητας. Επίσης οι παρεμβάσεις όσον αφορά την υγεία δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπονομεύουν την ε, προστασία υγείας στα βάλα των ομάδων του πληθυσμού. Υπό το πρίσμα των γενικότερων θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου, αναφέρεται στη μελέτη ότι τα δικαιώματα των ανθρώπων πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο τη διαδικασία λήψη αποφάσεων και όλοι οι σχετικοί νόμοι και οι αποφάσει και τα μέτρα πρέπει να βασίζονται στα πρότυπα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Η κυρία Κίρτον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για αυτές τις δύο παρουσιάσεις που νομίζω ότι έθεσαν πολύ σαφώς το πλαίσιο εντός του οποίου τίθενται και οι αναφορές που έχουμε λάβει. Δηλαδή οι πολιτικές επιλογές έχουν αντίκτυπο στους ασθενείς. Πολύ καλά θέσατε το πλαίσιο και καταλήξατε με κάποιες συστάσεις ε, για το τι πρέπει να κάνουμε. Η πολιτική υγεία είναι σε μεγάλο βαθμό εθνική αρμοδιότητα των κρατών μελών, η οργάνωση των συστημάτων υγείας. Υπάρχει κάποιο περιθώριο για παρέμβαση τον Ευρωπαϊκό Θεσμό Συνεργασία, τα θέματα δημόσιας υγείας, αλλά πολλά από τα διαφορετικά θέματα είναι εθνική αρμοδιότητα. Κάτι που θεωρώ πολύ ενδιαφέρον, εξετάζοντα ε, τις διάφορες εργασίες, είναι το παράδειγμα της Ολλανδίας και του Βελγίου που αγοράζουν από κοινού φάρμακα στα πλαίσια μιας προσπάθειας ε, επίτευξης καλύτερης ε, τιμής, δηλαδή περισσότερη αποτελεσματικότητα. Κάτι τέτοιο θα μπορούσαμε να το προωθήσουμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πώς συνεργάζονται οι χώρες, χωρίς κατά ανάγκη να εκχωρούμε περισσότερες αρμοδιότητες στην Ένωση, αλλά αν υπάρχει καλύτερο συντονισμός. Είναι κάτι που το έχετε εξετάσει. Υπάρχουν άλλα παραδείγματα τέτοιων πρακτικών. Αλλά το θετικό θέμα είναι ότι πρώτα απ' όλα ε, δείξατε πόσο έδειξε τους απλούς ανθρώπους στην κοινωνία μας και ιδίως τους πιο ευάλωτους ε, η λιτότητα. Η λιτότητα κυρίως έδειξε τις πιο μειονεκτικές περιοχές και τις πιο ευάλωτες ομάδες. Και αυτό το βλέπω εγώ και στην εκλογική μου περιφέρεια. Υπάρχουν τρομερές ανισότητες σε θέματα δημόσιας υγείας, οι οποίες οξύνονται όλο και περισσότερο. Ποιες θα ήταν οι τρεις βασικές σας προτάσεις για να αντιστρέψουμε αυτή την τάση, για να αντιμετωπίσουμε τα θέματα ανισοτήτων και προώθησης ενός εναλλακτικού θεματολογίου. Είναι απλώς θέμα δημόσιας χρηματοδότησης. Υπάρχουν και άλλα μέτρα που θα μπορούσαμε να προτείνουμε ούτω ώστε να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε τη ζωή των συμπολιτών μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Πρώτον για το Βέλγιο. Δεν έγραψα την έκθεση για το Βέλγιο εγώ, οπότε δεν έχω βαθιά γνώση του θέματος αλλά νομίζω ότι είναι πολύ καλό παράδειγμα το γεγονός ότι το Βέλγιο δεν περιέκοψε τις δαπάνες υγείας αλλά αλλά Πρώτα απ' όλα απαγόρευσε συμπληρώματα πληρωμών εάν οι ασθενείς ήταν σε δωμάτιο δίκλινο ή με περισσότερες κλίνες. Και αν ε, θέλετε να μου στείλετε περισσότερες ερωτήσεις, θα τις προωθήσω στον ε, συνάδελφο που έκανε την έκθεση για το Βέλγιο. Τώρα οι επιπτώσεις στα φτωχότερα και πιο ευάλωτα τμήματα των κοινωνιών μας Βεβαίως αυτό το διαπιστώσαμε σε όλα τα κράτη-μέλη. Και τι μπορεί να γίνει γι' αυτό. Βεβαίως πρέπει να αυξηθεί η δημόσια χρηματοδότηση του συστήματος υγείας ούτως ώστε αυτά τα ευάλωτα τμήματα του πληθυσμού να έχουν ένα ελάχιστο επίπεδο προστασίας, το απαιτούμενο σε ένα σύστημα υγείας. Και επίσης προτείνω να λαμβάνονται υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών όταν λαμβάνονται αποφάσεις για τον κλάδο της υγείας για να αποφύγουμε αυτές τις επιπτώσεις στα πιο ευάλωτα τμήματα. Η κυρία Πιτέλα. Ευχαριστώ πολύ πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ακούσαμε, αλλά έχω κάποιες αμφιβολίες. Τα προβλήματα του συστήματος υγείας δεν είναι πάντα θέματα χρηματοδότησης. Δεν είναι μόνο η ανεπάρκεια πιστώσεων που περιορίζει την πρόσβαση στην υγεία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε και μία έκθεση για την διαφθορά στον τομέα της υγείας στα 28 κράτη-μέλη και για τη διαφθορά γενικά και διαπιστώσανε ότι όσον αφορά τις δημόσιες προμήθειες ο τομέας της υγείας είναι εκείνος όπου παρατηρείται η περισσότερη διαφθορά. Και η διαφθορά έχει να κάνει με το γεγονός ότι πολλές φορές ζητούνται πληρωμές από τους ασθενείς για να πηδήξουν τους καταλόγους αναμονής για διάφορες θεραπείες. Για παράδειγμα, πολλές φορές ε, διάφοροι γιατροί προτείνουν και εκτελούν διάφορες ε, θεραπείες ή διάφορες επεμβάσεις που δεν είναι αναγκαίες. Αγοράζονται πολλές φορές ε, μηχανήματα που δεν χρειάζονται. Γιατί για παράδειγμα αν ένα νοσοκομείο δεν έχει συγκεκριμένη εξειδίκευση δεν χρειάζεται πολλές φορές τον εξοπλισμό που αγοράζει γιατί δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Οι διάφορες φαρμακευτικές εταιρείες κάνουν δώρα στους γιατρούς, ε, τους χαρίζουν ταξίδια, ούτως ώστε να συνταγογραφούν τα φάρμακα των εταιριών αυτών. Υπάρχουν πολλά φαινόμενα διαφθοράς. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι τα συστήματα υγείας ορισμένα κράτη-μέλη δεν είναι επαρκώς έντιμα και μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι υπάρχει μεγάλο ε, ε, ε, επιπλέον κόστος. Αυτό σημαίνει ότι όσο και αν αυξήσει τη χρηματοδότηση του συστήματος υγείας δεν βελτιώνεται η ποιότητα των υπηρεσιών λόγω ακριβώς αυτής της διαφθοράς. Πριν μιλήσουμε λοιπόν για το θέμα της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, πρέπει πρώτα απ' όλα να θέσουμε αυτό το ερώτημα. Τα συστήματα υγείας είναι βιώσιμα, είναι σωστά οργανωμένα. Διάβασα την έκθεση για την Ελλάδα για παράδειγμα. Και εκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει ότι είναι μεγάλη η διαφθορά στον τομέα της υγείας ε, στην Ελλάδα και αποτιμάται σε 33 δις το κόστος από τη διαφθορά. 33 δις. Άρα το μόνο πρόβλημα δεν είναι η αύξηση των πόρων. Δεν οδηγεί απευθείας σε αύξηση της ε, ποιότητας των υπηρεσιών υγείας ή αν θέλετε να το πω αντίστροφα η περικοπή των πιστώσεων υγείας δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι επιδεινώνεται η υγεία. Το πρόβλημα είναι ότι ένα μεγάλο ποσοστό της χρηματοδότησης της υγείας Πάει στραβά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να γίνουν πολλές ερωτήσεις και μετά να απαντήσετε συνολικά. Γιατί αλλιώς θα αργήσουμε πολύ. Παρακαλώ, κύριος για Να συμπληρώσω αυτά που είπε η συνάδελφός μου. Σωστά είπατε ότι η πρόσβαση στην υγεία είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Σίγουρα, συμφωνούμε όλοι. Όμως αυτά είναι κάτι που τα ακούμε κάθε μέρα. Εγώ πέρασα σε σοσιαλιστικό καθεστώς τα πρώτα 30 χρόνια της ζωής μου και λέγανε ότι ο καθένας έχει δικαίωμα στην υγεία και ήταν δωρεάν. Όμως υπήρχε πρόβλημα κόστους και η κοινωνία δεν ήθελε να το καταλάβει τότε. Γιατί τότε η λαοκρατική Γερμανία στην οποία ζούσα δεν μπορούσε να αγοράζει ε, επαρκή εξοπλισμό και γι' αυτό πέθαιναν οι άνθρωποι. Βεβαίω ε, ήταν δωρεάν το σύστημα, αλλά το σύστημα ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικό και δεν μπορούσε να παρέχει τι υπηρεσίε υγεία. Γι' αυτό συμπληρώνω. Βεβαίω, πολύ σωστά κάνατε αυτέ τι επιστημονικέ μελέτε, αλλά δεν θα έπρεπε. Πώ να το πω τώρα να ληφθεί υπόψη και η ανάγκη αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας. Δεν θα έπρεπε αυτό να συνδυάζεται με το ανθρώπινο δικαίωμα. Θα έπρεπε να είναι υποχρεωτική η σωστή λειτουργία του συστήματος υγείας. Στην Ευρώπη το βασικό είναι να μαθαίνουμε ένας από τον άλλον. Ο καθένας μας θεωρεί ότι το σύστημα υγείας του είναι άψογο Άρα δεν θέλει να ακούσει τι έχει να του πει κάποιος από την διπλανή χώρα. Όμως το θέμα τίθεται. Ποια ακριβώς είναι τα πρότυπα τα οποία πρέπει να ακολουθεί ένα σωστό σύστημα υγείας. Βεβαίως, ο καθένας πρέπει να έχει πρόσβαση. Αλλά οι πόροι είναι περιορισμένοι. Και επιπλέον, οι δυνατότητες που μας προσφέρει η σύγχρονη ιατρική είναι απεριόριστες και τίθεται και ερωτήματα ηθικής. Ήρθε ένας χειρουργός και μου είπε ότι βεβαίως αν δεν έχουμε άλλη λύση έχουμε και ένα σύστημα μεταμοσχεύσεων. Αλλά, μου είπε, έκανα μεταμόσχευση ενός ύπατος Όλοι ήταν ε, ικανοποιημένοι. Πήραμε το ύπαρ από ένα νέο ο οποίος πέθανε σε ένα τύχημα. Αλλά ήξερα ότι πολύ ε, σύντομα θα απορριφθεί. Και η απόφαση που πήρα ήταν ότι πρέπει αυτή η, αυτό το ύπαρ να μεταμοσχευθεί σε κάποιο νέο και κανένας ε, γυρότερος θα έπρεπε να πεθάνει. Βεβαίως, γιατί αναφέρω, αναφέρω τόσο ακραίο παράδειγμα διότι οι πόροι μας είναι περιορισμένοι από πολλές απόψεις. Άρα πρέπει να λειτουργούμε αποδοτικά και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να περιορίσουμε και την διαφορά. Να μην θεωρήσουμε ότι μπορούμε να τα κάνουμε όλα, ότι όλοι θέλουμε μόνο το καλύτερο και πάντα μπορούμε να έχουμε το καλύτερο για όλους τους ασθενείς. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι πρέπει να διερευνηθεί περισσότερο αυτό το θέμα που ανέφερα. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μπεθέρα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για την διοργάνωση αυτής της ε, ομάδας εργασίας. Πολύ βασικό να λάβουμε υπόψη ε, λοιπόν, τι έλεγα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι πολίτες σε αυτή την ανάλυση της κρίσης. γιατί έχουν επιπτώσεις όχι μόνο οι περικοπές λόγω της κρίσης, αλλά πρέπει να δούμε και τι πρόσβαση έχουν οι ασθενείς και στα φάρμακα και στις νέες τεχνολογίες. Πώς πρέπει να χορηγούνται οι άδειες στα νέα προϊόντα. Για την πρόσβαση στο σύστημα υγείας υπάρχουν πολλές χώρες που έχουν περικόψει κατά πολύ τους προϋπολογισμούς τους. Η Ισπανία η χώρα μου είναι μία από αυτές έχει κάνει από τις μεγαλύτερες περικοπές στην υγεία. Μεταξύ του 9 και του 13 μειώθηκε 16% η χρηματοδότηση υγείας, 10 δις δηλαδή περικόπησαν. Αυτό είχε πολλές επιπτώσεις και στην ε, αύξηση του χρόνου αναμονής και στην αντιμετώπιση των χρονίων ασθενειών και στην καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Αλλά θέλω να τονίσω κάτι που πρέπει να διευκρινίσουμε πολύ περισσότερο είναι οι επιπτώσεις ε, στα παιδιά. Είναι προφανές ότι η αύξηση της παιδικής ανεχίας θα έχει επιπτώσεις στην ε, υπόλοιπη ζωή των παιδιών, στην υγεία τους. Τα παιδιά στην Ισπανία ε, ζουν σε χειρότερη κατάσταση από το 2008 που ξεκίνησε η κρίση και αυτό σημαίνει ότι τα εγγυημένα δικαιώματα στην υγεία των πολιτών αυτών θίγονται και πρέπει να τους δοθεί προτεραιότητα. Γιατί έτσι μας υποχρεώνουν και οι διεθνείς συμβάσεις και οι ευρωπαϊκές συμβάσεις. Προφανώς και άλλα τμήματα του πληθυσμού είναι ευάλωτα, για παράδειγμα η άνω των 65 αλλά σε αυτή την πρώτη συζήτηση, επειδή θέλουμε να έχουμε και μια πολιτική προσέγγιση που είναι δουλειά μας να έχουμε, για να εγγυηθούμε την τήρηση των δικαιωμάτων των πολιτών, θα έπρεπε λοιπόν να λάβουμε υπόψη αυτή την ιδέα της ε, καθολικής κάλυψης ε, υγείας. Έτσι λέει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Όλοι οι πολίτες πρέπει να έχουν πρόσβαση σε επαρκή υγεία χωρίς να χρειάζεται να δαπανίσουν ένα μεγάλο τμήμα του εισοδήματό τους γι' αυτό και να πάσχουν κατά συνέπεια από ε, ανέχεια. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει πρόσβαση και στην περίθαλψη και στις ε, θεμελιώδεις τεχνολογίες και στα αναγκαία φάρμακα. Αυτό πρέπει να το δούμε σε σχέση με τις άδειες για τα φάρμακα και επίσης ε, το προσωπικό πρέπει να είναι επαρκώς καταρτισμένο. Καταλήγοντας λοιπόν, πιστεύω ότι θα έπρεπε να έχουμε ένα κατάλληλο, κάποιον οδηγό, τουλάχιστον να διευκρινίσουμε τι εννοούμε όταν λέμε ποιες είναι οι προτεραιότητές μας, ούτως ώστε η πρόσβαση των παιδιών στις υπηρεσίες υγείας να είναι εγγυημένη. Η συνάδελφος Ήβη. Ευχαριστώ. Έχω και εγώ μια ερώτηση. Ήθελα να μου πείτε πρώτα απ' όλα να πω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και μας ε, δημιουργεί πολλή σκέψη η παρουσίασή σας. Ε, πέραν των επιστημονικών στοιχείων που αποδεικνύουν τις επιπτώσεις των πολιτικών λιτότητας στην υγεία, όπως γνωρίζουμε όλοι στην Ευρώπη, πέραν αυτών, θεωρείτε ότι η υπογραφή εμπορικών συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών όπω η TTIP που βρίσκεται σε βάση διαπραγματεύση θα μπορούσε κατά κάποιο τρόπο να επηρεάσει και την υγεία όσον αφορά τη τιμή των φαρμάκων ας πούμε ή τα διπλώματα ευρεσιτεχνία ή την πρόσβαση στις υπηρεσίες πώς πιστεύετε ότι θα μπορούσε να επηρεάσει την υγεία των πολιτών διότι φυσικά είναι υπάρχει ευρία ανησυχία σε μεγάλο τμήμα του πληθυσμού. Ωραία να περάσω. Ωραία να απαντήσεις. Θέλω να πω ότι για τα φάρμακα ίσως περισσότερο να ασχοληθούμε μετά τις επόμενες παρουσιάσεις γιατί ιδιαίτερα ο κύριος Λαμάτα θα επιχειρήσει να απαντήσει όλα τα θέματα που τίθενται. Όπως για παράδειγμα το θέμα της οργάνωσης του συστήματος υγείας που κυρία Πιτέρα, μια μελέτη για την αποτελεσματικότητα και για την κάλυψη, την καθολική κάλυψη του πληθυσμού και η κυρία Μπεθέρα αναφέρθηκε στο μέλλον εφόσον αναφέρθηκε στο θέμα των παιδιών. Να κάνω κι εγώ όμως μία ερώτηση γιατί τίτλος ήταν τι μπορούμε να κάνουμε από πολιτική άποψη και η κυρία Ντάλη έκλεισε την ομιλία της αναφερόμενη σε θέματα που είναι θέματα πολιτικής εγγύηση της καθολικής πρόσβασης, την ισότητα, την ποιότητα και άλλα που μπορούμε να πούμε ότι αφορά τις, ε, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα το, συμβόλιο, το Συμβούλιο είπε ότι πρέπει να υπάρχουν ορισμένε αρχές και αξίες ότι πρέπει όλα τα κράτη-μέλη να τηρούν αρχές στην ε, πολιτική υγεία, για παράδειγμα, λοιπόν, καθολική πρόσβαση, αλληλεγγύη, ισότητα και πρόσβαση λοιπόν για όλους. Υπήρξε απόφαση λοιπόν που έχει να κάνει, υπήρξαν μάλλον αποφάσεις που βέβαια σχετίζονται με την ε, οικονομική συγκυρία, αλλά νομίζω ότι η βασική αρχή είναι η καθολικότητα της πρόσβασης. Βεβαίως πολλοί ομιλητές μίλησαν για το κόστος. Θέλουμε να εγγυηθούμε το θεμελιώδες δικαίωμα για όλους. Αλλά πολλές φορές τα θεσμικά όργανα αντιλαμβάνονται ότι σχετίζεται με την οικονομία. Και φυσικά πρέπει να μιλήσουμε για την ε, οικονομική διάσταση του θέματος. Αλλά το θέμα αυτό αφορά την ευημερία γενικά των ατόμων και την ποιότητα ζωής τους ή τις επιπτώσεις που θα έχει η έλλειψη υγείας, το βιωτικό επίπεδο, η, η παραγωγικότητά τους, όλα αυτά έχουν και οικονομική επίπτωση. Άρα η πολιτική υγείας έχει ευρύτερη οικονομική επίπτωση. Και αυτή είναι η ερώτησή μου. Δεν θα πρέπει να περιμένουμε ότι η καλύτερη υγεία θα έχει και θετικές οικονομικές επιπτώσεις. Δηλαδή και από οικονομική άποψη θα ήταν θετικό να δώσουμε περισσότερα για την υγεία. Πιστεύω λοιπόν πως θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε την άποψή σας και γι' αυτό. Γιατί πρέπει νομίζω να καταλήξουμε σε μια συνένεση. Να πούμε ότι η εγγύηση της καθολικότητας πρόσβασης θα έχει οικονομική επίπτωση. Πολύ πρόσφατα η Υπηρεσία για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα δημοσίευσε μια έκθεση πολύ ενδιαφέρουσα, όπου αναφερόταν στι οικονομικέ επιπτώσει του αποκλεισμού από, τους, από τα συστήματα υγείας των μεταναστών. Αυτό είπαν ότι θα είχε επιπτώσεις, ότι θα ήταν αναποτελεσματικό να τους βγάλουμε, ότι οικονομικά θα ήταν πιο αποτελεσματικό να συμπεριλαμβάνονται στην πρόσβαση στην υγεία. Θα ήθελα λοιπόν να μα πείτε ποιε είναι οι επιπτώσεις από οικονομική άποψη των περικοπών που γίνονται τώρα. Να δούμε λοιπόν τι σχέση η οικονομική κατάσταση στην υγεία. Τώρα δεν ξέρω πω θέλετε να απαντήσετε, αλλά όπως προτιμάτε. Thank you, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχετε υλικό για πολλά ακόμα εργαστήρια για τον οικονομικό αντικτύπο. Προσπαθούμε να το κάνουμε να το κατανοήσουν οι πολιτικοί ηγέτης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν έχουμε πετύχει και πολλά όμως. Δύο πράγματα όσον αφορά τις τεθήσεις ερωτήσεις. Δεν είμαι εμπειρογνώμων σε πολλούς από τους τομείς που εφήγησα. Για τις εμπορικέ συμφωνίες υπάρχει περιθώριο αυτές οι μεγάλες αυτές συμφωνίες, κυρίως αυτές που περιέχουν διατάξεις ευθέτηση διαφορών να έχουν αρνητικότατες συνέπειες για τα συστήματα υγείας και τους διάφορες παράγοντες για την υγεία σε σχέση με κοινωνικά ζητήματα. Έχω και εγώ γράψει ε, σχετικά ένα άθρο με συνάδελφο για την γενική δημοσιογεία. Το ερώτημα του Κέρτον Ντάρλινγκ για τρεις αρχές. Θα αναφερθώ σε μία από αυτές. Και ίσως σας κουράζω. Η, δημόσια χρηματοδότηση αφορά τη δημόσια υγεία άμεσα. Ο Ευρωβουλευτής έκανε μια ερώτηση για την υγεία των παιδιών και εύγλωτα το έθεσε το ζήτημα. Στις χώρες ΩΣΑ με υψηλό εισόδημα έχουμε τετραπλάσια διαφορά όσον αφορά τις συνέπειες που έχει η φτώχεια των παιδιών στον τομέα αυτό. Έχουν επιλογή ε, οι κυβερνήσεις για τη μετώπιση του προβλήματος ακολουθούν διαφορετικές προσεγγίσεις και υπάρχουν σχετικές ε, επιπτώσεις για τη δημόσια υγεία ανάλογα με τις ηλιμένες αποφάσεις. Όσον αφορά την πρώτη ερώτηση για τη διαφθορά στα συστήματα υγείας, υπάρχει πολλή διαφθορά, κυρίως στο ελληνικό σύστημα υγείας. Τεράστιο πρόβλημα όσον αφορά την πρόσβαση στο σύστημα υγείας στην Ελλάδα. Για να καταπολεμηθεί αυτό, τα συστήματα υγείας πρέπει να ελέγχονται προσεκτικότερα από τους αρμοδίους φορείς των κρατών μελών και θα πρέπει να θεσπιστούν και κυρώσεις. Αν διαπιστώνεται διαφθόρα, θα πρέπει να επιβάλλονται πρόστιμα, Φερρυπίν, ή αυστηρότερες κυρώσεις. Για να καταπολεμηθεί το φαινόμενο αυτό, και για να βελτιωθεί η πρόσβαση στην υγεία στην Ελλάδα, σε συστήματα υγείας. Πιστεύω ότι υπάρχει μια ανεπάρκεια στα συστήματα υγείας, περίθαλψης σε πολλά κράτη-μέλη και θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο παράγων των δημοσίων επενδύσεων αλλά πρέπει να γίνουν αποτελεσματικότερα συστήματα υγεία. Το 2005 στην Ιρλανδία Φερρυπίν κάποιος αρμόδιος του συστήματος υγείας εποπτικός φορέας έχει δημιουργηθεί. Έγιναν αλλαγές στο προσωπικό, στη δίκηση, πολλές αλλαγές που τελικά ήταν αρνητικές για την πρόσβαση στα συστήματα υγείας, αντί να επιλύσει προβλήματα. Πολλοί γιατροί και νοσηλευτές έχουν περισσότερα τα πετούμενα προσόντα στην Ιρλανδία και μεταναστεύουν, πάνε στο εξωτερικό, γιατί πληρώνονται καλύτερα και πηγαίνουν σε καλύτερα συστήματα υγείας. Ε, άρα χρειάζεται να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα των συστημάτων προνοίας για να καταπολεμήσουμε και τη διαφθορά και να, επίσης να επενδύονται και περισσότερα χρήματα από πλευράς ε, κυβερνήσεως. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ενδιαφέροντα. Οπότε, επειδή έχουμε κάποια καθυστέρηση, και θα μιλήσουν άλλοι τρει. θα περάσουν στο δεύτερο τμήμα να καταλήξουμε σε προτάσει για να αντιμετωπίσουμε τι προκλήσει που αντιμετωπίζουμε τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη πρώτον θα πάρει το λόγο ο κύριος Φερνάντο Λαμάντα που είναι ένας από αυτούς που συνέταξαν ε, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την έκθεση πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και θα μα μιλήσει για την οικονομική κρίση και την πρόσβαση στα ε, φάρμακα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριο Λαμάτα. Είναι τιμή η συμμετοχή σε αυτήν την τόσο σημαντική συζήτηση. Έχουμε ένα πρόβλημα, όπως ε, είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, το οποίο είναι ότι στην Ευρώπη, στα διάφορα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Υπάρχει ένα πραγματικό πρόβλημα πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας. Θεωρούμε ότι 18 εκατομμύρια δεν έχουν δυνατότητα πρόσβασης στις ε, υπηρεσίες υγείας που δικαιούνται. Άρα σε χώρες με υψηλό ε, και μέσο επίπεδο εισοδήματος ε, υπάρχει αυτό και είναι απαράδεκτο. Και γιατί συμβαίνει. Θα ασχοληθώ με δύο θέματα. Πρώτον, οι περικοπέ των δημοσίων ε, χρηματοδοτήσεων, ήδη αναφέρθηκε. Και δεύτερον, η υψηλή τιμή των νέων φαρμάκων, που επίσης ε, αποτελούν ε, φραγμό στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. ήδη μεταξύ 2008 και 2013 στην... σε πάνω από τα μισά κράτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση μειώθηκαν οι προπολογισμοί Και αυτό σήμαινε ότι αυξήθηκε η συμμετοχή των ασθενών, μειώθηκε η χρηματοδότηση κάποιων φαρμάκων και ως ε, συνέπεια της μη πρόσβασης ε, κάποιων ομάδων του πληθυσμού δεν έχουν πρόσβαση και σε φάρμακα. Γιατί έγιναν αυτές οι περικοπές. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Το σημαντικό δεν είναι μόνο να δούμε την επίπτωση ότι μειώθηκαν ε, πάνω από 45 δις των προϋπολογισμών. Αλλά παράλληλα τα κράτη-μέλη έδιναν ένα μεγάλο τμήμα των προϋπολογισμών τους πάνω από ένα τρισεκατομμύριο ευρώ πήγε στην αναχρηματοδότηση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Και επίσης έγινε και, έγιναν και δανειδοτήσεις από την Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, επίσης ενός 3 εκατομμυρίου ευρώ και παράλληλα, και αυτό δεν είναι επίπτωση της κρίσης, αλλά επιδεινώθηκε κατά την κρίση στις χώρες της Ένωσης αυξήθηκε κατά πολύ η φοροδιαφυγή που θεωρούν επίσης οι υπηρεσίες της Κομισιόν ότι είναι του ύψους ενός τρεις. Άρα όταν λέμε ότι πρέπει να εγγυθούμε την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας πρέπει να μιλήσουμε επίσης για καλύτερη ρύθμιση του χρηματοδοτικού τομέα, κατά καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση ενός ε, σταδιακού συστήματος φορολόγησης. Δηλαδή μια νέα ισορροπία μεταξύ του χρηματοπιστωτικού τομέα και της υπόλοιπης κοινωνίας. Γιατί είναι τόσο υψηλέ οι τιμές των νέων φαρμάκων. Και εδώ παρατηρούμε μια ανισορροπία. Δεν υπάρχει μια λογική σχέση. Οι πολύ υψηλέ τιμές των νέων φαρμάκων παρεμποδίζουν ή καθυστερούν την πρόσβαση πολλών ασθενών στις αναγκαίες θεραπείες και αφαιρούν του αναγκαίου πόρου για να αντιμετωπιστούν άλλα προβλήματα υγεία εκατομμυρίων ατόμων και θέτουν κινδύνο την βιωσιμότητα των συστημάτων περίθαλψη. Λογικά οι επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα προσπαθούν να θέσουν το πιο υψηλό τίμημα που μπορούν να πληρώσουν οι αγορές, δηλαδή τα συστήματα υγείας ή ασθενείς. Εάν υπήρχε ανταγωνισμός θα μπορούσαν να μειωθούν οι τιμές. Αλλά στις δεκαετίες 60 και 70 τα κοινοβούλια και οι κυβερνήσεις ενέκριναν τις άδειε των φαρμάκων για να προστατεύσουν τις καινοτόμες επιχειρήσεις. Τους έδωσαν λοιπόν μονοπόλιο, την αποκλειστική ε, είσοδο στην αγορά δηλαδή, των φαρμάκων αυτών. Αυτό το μονοπόλιο ισχύει για 20 χρόνια για να μπορέσουν να καλύψουν το κόστο τη έρευνα. Αυτή είναι και όχι καμία άλλη η αιτιολόγηση του μονοπόλιου. Αλλά οι επιχειρήσει το χρησιμοποίησαν για να θέσουν πολύ υψηλέ τιμέ, Πολύ πάνω από το κόστο τη έρευνα για την ε, διαμόρφωσή του Και οι κυβερνήσει και τα κοινοβούλια το επέτρεψαν. Παράδειγμα, σύμφωνα με την έκθεση ενός... Ε, συγγνώμη, την έκθεση τη γερουσία των ΗΠΑ για την υπατήτητα ΣΕ, το συνολικό κόστο για ένα συγκεκριμένο φάρμακο ήταν 942 εκατομμύρια δολάρια. Οι πωλήσει των πρώτων 21 μηνών ήταν 26 δι, Δηλαδή πάνω από ένα δι το μήνα. Δηλαδή το κόστο τη έρευνα όχι μόνο καλύφθηκε, αλλά πολύ παραπάνω. Άρα το μονοπόλιο δεν δικαιολογείται πλέον. Θα έπρεπε να μειωθεί η τιμή, να πέσει στο κόστο παραγωγή ή να υποχρεωθεί η εταιρεία να δώσει άδεια στα κράτη να ε, παράγουν το προϊόν αυτό. Έτσι θα μπορούσαμε, εάν είχαμε αυτή τη δυνατότητα αυτού του φαρμάκου σε χαμηλή τιμή, να εξαλείψουμε αυτή την ασθένεια. Γιατί δεν γίνεται αυτό. Όπως είπαμε, το κόστος της έρευνας δεν αιτιολογεί τόσο υψηλές τιμές. Όταν το είπαμε αυτό, τότε είπαν ότι έχει ένα συγκεκριμένο, συγγνώμη, μια συγκεκριμένη τιμή αυτό το προϊόν λόγω της αξίας που έχει διότι μπορεί να αυξήσει την ε, ζωή και τα λοιπά των ασθενών. Αλλά καμία από αυτές ε, τις αιτιολογίες δεν μπορεί να δικαιολογήσει το φαινόμενο. Ένα άλλο φαινόμενο για την αύξηση των τιμών είναι ότι έχουν γίνει χρηματοπιστωτικό προϊόν τα φάρμακα. Οι υψηλέ τιμέ αυξάνουν τι τιμέ, βεβαίω. Αλλά παράλληλα αυτό σημαίνει ότι είναι ένα μήνυμα προ τι κεφαλαγορέ που αξιοποιείται για να αυξηθεί η τιμή των μετοχών των εταιρεών αυτών. Αυτά που κερδίζουν οι εταιρείε αυτέ στο χρηματιστήριο και οι τα διευθυντικά τους ε, στελέχη σημαίνει ότι χρησιμοποιείται το φάρμακο ως χρηματοπιστωτικό προϊόν. Του εξήγησαν διάφορες ε, εργασίες του Μάρτιν Χρέλ για τα φάρμακα Τούριν και Καλοβίος. Πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι αυτός ο τρόπος χρηματοδότησης είναι επιπλέον αναποτελεσματικός. Το είπαν και ορισμένοι κοινοβουλευτικοί ότι θέλουμε περισσότερη αποτελεσματικότητα δεν είναι αποδοτικό για το σύνολο τη κοινωνία αυτό το σύστημα. Είναι πολύ αποτελεσματικό για τι φαρμακευτικέ εταιρείε, αλλά καθόλου για την κοινωνία που χρηματοδοτεί αυτό το μοντέλο. Το υπερβολικό κόστο συντα... συνταγογράφησης, τα... οι παρενέργειες που θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί, που η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι είναι γύρω στα 80 δις, το υπερβολικό κόστο τη διαφήμιση και του μάρκετινγκ, και το ποσοστό κέρδους που είναι πάνω από διπλό από άλλους κλάδους σημαίνει πως αυτό το είδος χρηματοδότησης της έρευνας είναι αναποτελεσματικό. Θα πρέπει να έχουμε ένα άλλο μοντέλο. Θα πρέπει να χρηματοδοτείται απευθείας η έρευνα. Θα είχαμε μια μείωση 30% του κόστους για τα φάρμακα έτσι. Δηλαδή θα είχαμε κάθε έτος εξοικονομήσει 80 δις και μήπως ε, αξιοποιήσαμε ε, με αυτόν τον τρόπο περισσότερο τις δυνατότητες ε, για καινοτόμα φάρμακα. Όμω διαπιστώσαμε ότι κάθε χρόνο πεθαίνουν 25.000 άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν υπάρχουν, επαρκή, συγγνώμη, δεν υπάρχουν αποτελεσματικά αντιβιωτικά. Επίσης αργούν να υπάρχουν ορισμένα φάρμακα σε κάποιε χώρε, γιατί κάποιε χώρε δεν μπορούν να πληρώσουν τι τιμέ που απαιτούν οι φαρμακευτικέ. Ορισμένα αποτελεσματικά αλλά φθηνά φάρμακα ε, αποσύρονται από την αγορά για να εισαχθούν άλλα πιο ε, ακριβά και σε ορισμένες ε, περιπτώσεις μάλιστα είναι το 75% των νοσοκομείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν λαμβάνουν ορισμένα φάρμακα. Επίσης ξέρουμε πολύ καλά ότι πολλές φορές διαστρεβλώνονται οι κλινικές δοκιμές, αυξάνονται οι κίνδυνοι για τους ασθενείς που συμμετέχουν στις κλινικές δοκιμές και δεν δημοσιεύονται αρκετά νωρί τα αποτελέσματα. Υπάρχει εναλλακτική δυνατότητα. Το 2010 το Συμβούλιο Υπουργών της Ένωσης ζήτησε να γίνει μια εξέταση τη δυνατότητα να διαχωριστεί η χρηματοδότηση τη έρευνα από το σύστημα καθορισμού των τιμών. Τότε αφορούσε χώρε ε, χαμηλού εισοδήματο. αλλά τώρα αφορά όλες τις χώρες Ευρώπη. Γιατί ούτε πια οι χώρες Ευρώπη δεν μπορούν να πληρώσουν το κόστο των νέων φαρμάκων. Θα έπρεπε να έχουμε μια πλατφόρμα δημόσια χρηματοδότηση τη έρευνα όπου θα υπήρχε συντονισμό θα ήταν ανοιχτή η έρευνα, δηλαδή πρόσβαση στα αποτελέσματα και τα φάρμακα θα απολούνται στην τιμή του γενοσύμου. Και τι μέτρα μπορούμε όσο εξετάζεται αυτή τη δυνατότητα να υιοθετήσουμε πιο ε, βράχη πρόθεσμα. Βεβαίω, λόγω της κρίσης είχαμε τα θετικά μέτρα, όπως για παράδειγμα πιο αυστηρή αποτίμηση των αποτελεσμάτων της δημόσιας χρηματοδότησης των εφαρμάκων, η μείωση των περιθωρίων κέρδους, κέρδους των εταιριών, η κοινή αγορά ε, φαρμάκων των χωρών Benelux ήδη αναφέρθηκε, η αύξηση της χρήσης των γενοσύμων, βελτίωση της ε, συνταγογράφησης, βελτίωση της χορήγησης των φαρμάκων ή η χρήση πιο φθηνών φαρμάκων. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε ως θεσμικά όργανα της Ένωσης. Μερικές ιδέες. Μεταξύ αυτών να δημιουργήσουμε μια επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μελετήσει το κόστος και τις τιμές των φαρμάκων διότι μόνο μέσω γνώσης και διαφάνειας μπορούμε να αλλάξουμε την κατάσταση. Επίσης θα μπορούσαμε να διαπραγματευτούμε τιμές που να βασίζονται στο κόστος της κατασκευής και της έρευνας και ένα αντιλογισμένο κόστος. Ε, στο μέσο όρο του ποσοστού κέρδους ε, παρόμοιων κλάδων. Και επίσης θα μπορούσαμε να αποφύγουμε τις μονοπωλιακές καταστάσεις. Οπότε θα υπήρχε περισσότερο περισσότερος ανταγωνισμός. Επίσης θα πρέπει να χρηματοδοτήσουμε την Ευρωπαϊκή, ε, τον Ευρωπαϊκό Φορέα Φαρμάκων και άλλους ε, εθνικούς φορείς να καταρτήσουμε καλύτερα ε, το νοσηλευτικό προσωπικό και να βοηθήσουμε και τις ενώσεις ασθενών, όλα αυτά πρέπει να είναι ανεξάρτητα από τη φαρμακευτική βιομηχανία, να ελέγχουμε τις συγκρούσεις συμφερόντων. Και επίσης θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε μια σφαιρική πλατφόρμα για την έρευνα. Αυτό μπορεί να ξεκινήσει μέσω μιας πρωτοβουλίας για την έρευνα για τα αντιβιωτικά. Έχουμε την ευθύνη να αναλύσουμε τα προβλήματα αυτά λεπτομεριακά και να δώσουμε απαντήσεις. Είναι απαράδεκτο να υπάρχουν εκατομμύρια άτομα στην Ευρώπη και πολύ περισσότερα σε άλλα τμήματα του κόσμου που δεν έχουν πρόσβαση στα φάρμακα. Είναι απαράδεκτο να παραβιάζεται αυτό το δικαίωμα κάθε μέρα ενώ με άλλο τρόπο ε, χρηματοδότηση θα μπορούσαμε να το εγγυηθούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Λαμάτα για την καταπληκτική παρουσίασή σας. Να δώσουμε το λόγο τώρα στον κύριο Ρομπέρτο Μπερτολίνη, εκπρόσωπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Θα μιλήσει για την πρόσβαση στις ε, υπηρεσίες υγείας στις χώρες που έχουν φυγεί από την κρίση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε για την πρόσκληση να έρθω εδώ να παραστώ σε αυτό το άκρος ενδιαφέρον εργαστήριο, στην ενδιαφέρουσα συζήτηση. Καταρχάς θέλω να πω ότι δεν μπορώ να παρασυμφωνήσω με αυτά που είπε ο Δ. Σέκερ για το θέμα των ε, δημοσίων επενδύσεων για τον τομέα της δημόσιας υγείας και πώς επηρεάζεται. Θα ήθελα να προσθέσω και άλλη μια φράση προς υπόμνησή σας ότι η υγεία είναι πολιτική επιλογή. Αυτό πάντα υπερισπέζει υπερασπιζόμασταν επανειλημμένα. Οι, οι, διάφοροι, οι διάφορες συνιστώσεις και οι διάφορες συντελεστές επηρεάζονται από την επιλογή ή την έλλειψη επιλογών σε κάποιες περιπτώσεις. Λοιπόν, θα σας παρουσιάσω το όλο ιστορικό, το υπόβαθρο, θα είμαι λακωνικότατος, πολλά ήδη καλύφθηκαν. Στο δεύτερο τμήμα θα αναφερθώ σε κάποια μαθήματα τα οποία έχουμε αποκομίσει από τις εμπειρίες όπως αναφέρθηκε από τον Κόσμιο Οργανισμό Υγείας σε διάφορες περιστάσεις και τέλος θα καταλήξω σε κάποια συμπεράσματα. Τώρα, καταρχάς, όπως ήδη αποδείχθηκε από τον καθηγητή Σρέκα και από άλλους ε, ομιλητές του πάνελ, υπάρχουν σημαντικά στοιχεία σχετικά με την επιρροή των οικονομικών κλειδονισμών επί της υγείας. Πρώτα απ' όλα αυτά τα γεγονότα επηρεάζουν τους ενήλικες, το είδαμε και σε κάποιες περιπτώσεις και θετικές επιπτώσεις για τη μείωση των οδικών ατυχημάτων Φερρυπίν. Αλλά δεν επηρεάζουν τον καθένα με τον ίδιο τρόπο. Η υγεία επιδεινούται σε ανθρώπους που χάνουν τη δουλειά τους, που έχουν προβλήματα κοινωνικο-οικονομικά. Επίσης μάθαμε από τις πρώτερες εμπειρίες ότι οι αρνητικές συνέπειες μπορούν να μειωθούν, υπάρχουν σχετικές στρατηγικές. Κάποιος από τους ευρωβουλευτές αναφέραν κάποια θέματα προηγουμένως που ε, είναι σημαντικότατα. Επίσης υπάρχουν και αντικυκλικές κοινωνικο-οικονομικές δαπάνες. Για να αντισταχθεί κανείς της, ρο, της ροής του κύκλου για να προστατεύσει τους πλέον ευάλωτες από την οικονομική κρίση είναι ένα μέτρο και να προστατεύουμε την πρόσβαση στην ε, περίθαλψη. Είναι κρισίμου σημασίας κυρίως για εκείνους ανθρώπους που κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους ή ζουν στη φτώχεια. Οι προλαλήσαντες ήδη απέδειξαν, έδειξαν τα στοιχεία από την Ελλάδα. Αυτό είναι πρόσφατο έγγραφο για τη σχέση μεταξύ αυτοκτονίας και των συνθήκων. Να αναφέρω μια σκέψη εδώ. Εδώ η καμπύλη που βλέπετε πάνω δείχνει την αύξηση στις αυτοκτονίες και αντικατοπτρίζει ε, τους άρενες από 20 μέχρι 59 ε, και άρενες από 60 και πάνω. Αυτή είναι η ομάδα που έχει πληγεί περισσότερο από την κρίση και έγινε κάποια αξιολόγηση και κάθε ποσοστό παραπάνω 1% ε, ε, ε, οδηγεί σε μια αύξηση 0,19% στο, στο ποσοστό αυτοκτονιών. Ποιο είναι το πρώτο μάθημα. Οι εκείνοι που λαμβάνουν τι αποφάσει, οι πολιτικοί έχουν επιλογέ ακόμα και σε περίοδο λιτότητα. Πριν περικόψουν τι δαπάνε για την υγεία, θα πρέπει να δούνε και ποιο είναι το αντιστάθμισμα, ποια είναι η συνέπεια, τι κερδίζουμε, τι χάνουμε, κόστο όφελο. Επίση να εξισορροπήσουν οι ανάγκε οι βραχυπρόθεσμε και οι πανκροπρόθεσμες. Αυτό επιδείχνει σε μια κρίση. Όταν σταματά να παρέχεις ή δυσκολεύεσαι να δώσεις ε, ε, φάρμακα κατά ε, σηματιώσεως, παραδείγματος χάρη, και δημιουργούνται περιπλοκές και το κόστος ε, για το σύστημα υγείας τελικά είναι μεγαλύτερο από ό,τι θα ήταν αν μπορούσες να καλύπτες τους ανθρώπους με προστασία κατά κάποιων ασθενειών. Και αν περικοπούν οι περικοπές θα πρέπει να είναι ε, σωστά. Πρέπει να εξετάζονται τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα και δεν θα πρέπει να γίνονται πολλές οριζόντιες περικοπές. Θα πρέπει να σκέπτονται αυτοί πριν που παίρνουν τι αποφάσεις. Λοιπόν, η κυρία Κέλλη έκανε κάποιες παρουσιάσεις και έγινε κάποια συζήτηση και ακούστηκαν κάποια πράγματα και αναφορές σε κάποιες χώρες όπως είναι το Βέλγιο και η Ολλανδία που υιοθέτησαν κάποια αντικυκλικά μέτρα προσπαθώντας να προστατεύσουν κάποιες ομάδες του πληθυσμού και αυξάνοντας έτσι την αποδοτικότητα. Και αυτό συνέβη. Ε, βλέπουμε Βέλγιο και Ολλανδία στο αριστερό τμήμα της διαφάνειας. Βλέπουμε αύξηση των δημοσίων δαπανών κατά την περίοδο της κρίσης, παρόλο που οι κρίση ήταν λιγότερο σοβαρή σε κάποιες χώρες. Από την άλλη πλευρά βλέπετε από την άλλη πλευρά ότι οι χώρες ε, έλαβαν μέτρα που ακολουθούσαν τον κύκλο. Ε, μείωναν τους πόρους της επενδύσης στον τομέα της υγείας και αυτό πιστεύουμε ότι είναι κάτι αρνητικό σαν μέτρο. Δεν είναι θετική η προσέγγιση. Τώρα, το άλλο θέμα είναι ότι οι περικοπές και οι οικονομίες δεν είναι δεν έχουν τέτοια αποτελέσματα όσον αφορά την αποδοτικότητα. Αν δούμε από τη μία πλευρά την αποδοτικότητα και τις οικονομίες από την άλλη βλέπουμε την κατάσταση κατά την οποία μέσω σοφών επιλογών μπορείς να πετύχεις τα ίδια και περισσότερα με λιγότερους πόρους το τρόπος μπορείς να κάνεις οικονομίες και να αυξήσεις την αποδοτικότητα, η καλύτερος εφοδιασμός ε, μπορεί να επιτευχθεί, ε, να μην υπάρχουν πλεονάσματα στον φωτοδυναμικό, να γίνει περιορισμός των ανθρωπίνων πόρων, αν υπάρχει δυνατότητα, να μην, είναι, να μην υπάρχουν πολύ φουσκωμένοι μισθοί ε, όταν αυτό διαπιστωθεί. Υπάρχουν δυνατότητες λοιπόν να γίνουν ε, επενδύσεις και να κάνεις τα ίδια περισσότερα με λιγότερους ε, πόρους. Βέβαια, μπορείς να κάνεις και λέσα με, τους, με λιγότερους πόρους, αυτό είναι προφανές, αλλά μπορεί να αυξήσει την αναποτελεσματικότητα κάνοντας οικονομίες. Αν κάνεις περικοπές χωρίς να κάνεις αυτές τις επιλογές στις δημόσιες υπηρεσίες. Μειώνει τη διαθεσιμότητα των ε, γιατρών στην πρωτοβάθμια περίθαλψη ε, και τη, μειώνεις την πρόσβαση. Οπότε μπορούν να πηγαίνουν στις, ε, στα επίγοντα περιστατικά οι άνθρωποι για να καλύψουν τις ανάγκες τους, οι ασθενείς. Και αυτό μπορεί να είναι πολύ δαπανηρό σαν λύση. Άρα έχεις, φαίνεται σε να μειώνεις το κόστος, στην πραγματικότητα όμως τα αυξάνεις το κόστος. Διότι ε, πρέπει τα ε, πήγοντα περιστατικά να καλύπτουν προβλήματα που διαφορετικά θα μπορούσαν να καλυφθούν πιο φθηνά από τον ε, παθολόγο. πρέ μπορούμε να, να, κερδίσουμε σε απόδοση χωρίς μεγάλες οικονομίες, Τιώνοντας ε, τον έλεγχο των δαπανών μέσω σωστού σχεδιασμού, σωστής αξιολόγησης ε, ε της χρησιμοποιουμένης τεχνολογίας και να βελτιώσει την πρόληψη. Ε, θα το δούμε αργότερα αυτό το θέμα της, τι γίνεται με την πρόληψη στον τομέα της υγείας. Μπορείς επίσης να μειώσεις το κόστος και να αυξάνοντας την αποδοτικότητα κατά πολύ όταν δεν υπάρχουν σωστά εναλλακτικά μέτρα που να βελτιώνουν την απόδοση. Μπορεί να καταλήξει να αυξήσει το κόστος. Λοιπόν, το θέμα της δημόσιας υγείας, πώς να το πω, είναι μοιοπία, ένα είδος ασθένειας, μια μοιοπία που δείχνουν εκείνοι που διαμορφώνουν την πολιτική. Βλέπετε από τις διαφάνειες, οι μεγαλύτερες περικοπές στις χώρες που έχουν πληγεί από την κρίση, από το 2007 μέχρι το 2011, ε, έγινε στον τομέα της δημόσιας υγείας και της προλήψεως. Ε, και αυτό δεν είναι σωστή απόφαση. Διότι ο τρόπο μειώνει τη δυνατότητα να κάνει μεγάλε οικονομίε στο μέλλον μέσω προλήψεως εμφανίσεω ασθενειών. μειώνοντα την εμφάνιση των ασθενειών που συνδέονται φερρυπίν με τη διατροφή, με φυσική δραστηριότητα ή ε, εμβολιασμού. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να διορθωθεί, μπορεί να διορθωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ένα ρόλο να παίξουν σχετικά με αυτό. Ε, Πολλέ χώρε στην Ευρώπη έχουν μόνο 3% του προπολογισμού που διατίθεται για την πρόληψη και τη δημόσια υγεία και σε κάποιες χώρες αυτό το ποσοστό και αυτές είναι οι χώρες που έχουν ε, πληγεί περισσότερο από την κρίση αυτές, αυτό το ποσοστό λέγω που είναι, είναι κάτω από το 1% που αυτό είναι απαράδεκτο, γελίο θα έλεγα. Γι' αυτό πρέπει να εστιαστούμε λοιπόν στην αποδοτικότητα και είναι σημαντικό αυτό, αλλά έχει και τα όρια του αυτή η προσέγγιση, της ε, η προσέγγιση. Η βελτίωση της αποδοτικότητας, όπως ανέφερε και ο κύριος Γιάρ, πρέπει να είναι μόνιμη προσπάθεια, όχι μόνο μια προσπάθεια που καταβάλλεται κατά την περίοδο κρίσης και μόνο. Πολλές χώρες ε, αρκετά γρήγορα ε, έδρεψαν τους καρπούς που κρεμόταν χαμηλά στο δέντρο, παραδείγματος χάρη, ε, μείωσαν ε, τις τιμές από κάποια ακριβά φάρμακα. Αλλά χρειάστηκαν ε, και χρειάζονται περίπλοκες μεταρρυθμίσεις και αυτές πρέπει να στηρίζονται από δημιουργία δυναμικού, επενδύσεις και ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα και καμιά φορά η ανάγκη περικοπής και μείωσης του προϋπολογισμού πρόθεσμα, εμποδίζει την εισαγωγή μακροπροθέσμων μεταρρυθμίσεων και αυτό δημιουργεί κόστος μακροπρόθεσμα, συγγνώμη. Λοιπόν, τα κέρδη αποδοτικότητα δεν μπορούν να καλύψουν το μεγάλο κενό που υπάρχει μεταξύ εσόδων και δαπανών. Δεν υπάρχουν αρκετές περικοπές για να καλυφθεί αυτό το κενό. Τελικά, χρειάζεται ε, οικονομική προστασία και πρόσβαση στην περίθαλψη. Πρέπει να έχει προτεραιότητα, μάλλον δράση προστατευτική για τους πιο ευάλωτους. Καμιά φορά η προστασία που παρεσχέθη έφτασε πολύ αργά και ήταν χαμηλού επίπεδου, κυρίως για συνταξιούχους, φτωχούς συνταξιούχους τις στοχές ε, κοινωνικές ομάδες και η, δράση προστασίας δεν, δεν είχε προτεραιότητα στις διαδικασίες προσαρμογής που εξέταζαν μόνο τη μακροοικονομική εικόνα και αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη. Οι περικοπές των δαπανών μπορούν να εξίσου επιβλαβείς όπως και οι περιορισμοί κάλυψης όσον αφορά την οικονομική προστασία και πρόσβαση. Βραχυπρόθεσμα, παραδείγματος χάρη, μεγάλες και περικοπές σε προπολογισμούς για νοσοκομεία, παραδείγματος χάρη, αυξάνουν τον χρόνο αναμονής ε, και τα φακελάκια και αυτό βοηθά να αυξηθεί η διαφθορά. Πιο μακροπρόθεσμα οι περικοπές όσον αφορά το προσωπικό και η περικοπή των πληρωμών, κυρίως όταν είναι ήδη χαμηλή μισθή, μπορεί να έχει παρόμοιο αποτέλεσμα ε, και να οδηγήσει σε μετανάστευση των επαγγελματιών του τομέα και να πάνε σε άλλες χώρες όπου η αμοιβή είναι καλύτερη και συνεπώς έτσι ε, δημιουργείται ένα αποτέλεσμα αντίθετα από το ευκταίο Στι χώρε προέλευση εκεί που μεταναστεύουν. Και τώρα κλείνοντα, οι, οι ανάγκες που δεν καλύπτονται, τι σημαίνει αυτό. Ανάγκε υγεία που δεν καλύπτονται από το σύστημα υγεία λόγω ε, ε, διότι είναι μακριά ο τόπο περίθαλψης και οι δαπάνε υψηλέ. Εδώ από το 2009 και μετά, μέχρι το 2009 μειωνόταν, για τους στοχότερους κυρίως, αλλά το 2009 μέχρι το 2013 τι έγινε. Οι μη καλυπτώμενε ανάγκες παρέμεναν στα ίδια επίπεδα, σιγά σιγά αυξανόταν με την εξαίρεση βέβαια των ε, πιο πλουσίων 20%. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν αυτό να το λάβουμε ε, υπόψη για να το αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο. Λοιπόν, η μείωση των ανετικών συνεπειών της κρίσης απαιτεί πολύ καλή διακυβέρνηση, ηγεσία, ε, θα πρέπει να λαμβάνονται αποφάσεις λαμβάνοντας υπόψη τον περίπλοκο χαρακτήρα των ζητημάτων και ποιο είναι το αντιστάθμισμα, ποιο είναι το αποτέλεσμα. Ε, παρά την ευαισθητοποίηση, η πρόθεση ε, της πρόσβασης και της οικονομικής προστασίας δεν αποτελούσε προτεραιότητα σε προγράμματα οικονομικής προσαρμογής και αυτό θα πρέπει να καλυφθεί, να εξεταστεί προσεκτικότατα. Υπάρχουν περιορισμένα στοιχεία για τα αρνητικά αποτελέσματα Δείξαμε κάποια στοιχεία, αλλά έχουμε ενδείξει ότι ο αριθμό άλλων στοιχείων, άλλων γεγονότων συνέβαιναν λόγω τη κρίση, αλλά δεν είχαμε αρκετά γρήγορα τα στοιχεία στα χέρια μα για να σα δώσουμε αρκετέ πληροφορίε, για να σα πω τι έγινε πέρσι ή πρόπερσι. Άρα χρειάζεται καλύτερη παρακολούθηση και συλλογή στοιχείων, καλύτερη χρήση των ε, στοιχείων. Λοιπόν, η ανταπόκριση του στήματο υγεία είναι πάρα πολύ σημαντικό για να αντισταθμούν οι αρνητικέ συνέπειε οικονομική κρίση που πλήττει κυρίω του φτωχότερου αλλά βασική μοχλή είναι εκτός του συστήματος υγείας. Θα πρέπει οι υπεύθυνοι για θέματα υγείας και για τα θέματα οικονομικών να συνομιλήσουν και χρειάζεται διάλογος. Είναι μια δυνατότητα και ευκαιρία οι δύο τομείς να συνομιλήσουν, ο τομέας της υγείας και των οικονομικών και αυτός ο διάλογος δεν πιστεύω ότι λαμβάνει χώρα. Στο Κοινοβούλιο ζητάμε να υπάρχει συζήτηση με την Επιτροπή Προπολογισμών ή με τους ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι για τα οικονομικά θέματα και είναι πολύ δύσκολο για μας, για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και για άλλους ε, φορείς να έχουν ε, διάλογο με τους συναδέλφους και αυτό θα πρέπει να γίνει. Και επανέρχομαι στην αρχική πρόταση που ανέφερε ο καθηγητής Ρέκερ. Ε, είναι, είναι θέμα δημόσια υγείας η δημόσια χρηματοδότηση. Αν δεν μιλήσουμε με τους υπευθύνου όμως, αν δεν υπάρξει διάλογος, ε, μιλάμε με αυτούς που έχουν ήδη πιστεί. Πρέπει όμως να καλύψουμε αυτό το κενό και ενθαρρύνω τους παρόντες ευρωβουλευτές και εσάς κυρία Πρόεδρε να δημιουργήσετε αυτή τη δυνατότητα, να λάβετε μια πρωτοβουλία να καθίσουν και στο τραπέζι εκείνοι που ασχολούνται με τα οικονομικά και τον προπολογισμό και τη δημόσια υγεία και τους υπεύθυνους για κοινωνικά θέματα για να συνομιλήσουν. Θα είναι ένα μικρό βήμα προς καλύτερη συνεννόηση, ε, να καταλάβει ένας τον άλλον καλύτερα και να εξεταστούν οι κοινωνικές πτυχές που καμιά φορά αμελούνται. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μπερτολίνη <clears throat> και ελπίζω να μπορέσουμε να κάνουμε διάλογο με βάση αυτά που ακούστηκαν γιατί είναι πολύ σημαντικό. Και τώρα <clears throat> ο κύριος Καρβάλιο της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που θα μα μιλήσει για την σημερινή και μελλοντική κατάσταση της πολιτικής υγείας και της πρόσβαση σε περίθαλψη και φάρμακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρακαλώ. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Επιτροπή Αναφορών που δίνει στη, μας, ε, στην Επιτροπή τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε το θεματολόγιο για την πρόσβαση στην υγειονομική περιθαλψή. Προτιμώ πάντα να ξεκινώ με τον ορισμό της πρόσβασης ε, στην υγειονομική περιθέρωση. Τι εννοούμε δηλαδή. Γιατί ξέρετε πολύ συχνά το πρόβλημα είναι ότι ο κόσμος αναφέρεται σε κάτι διαφορετικό με αυτό τον όρο. Θα σας δώσω λοιπόν τον ορισμό που παρουσιάστηκε σε μια ανακοίνωση που υιοθέτησε η Κομισιόν το 2014. Πρόκειται για την ανακοίνωση για τα αποτελεσματικά προσβάσιμα και ανθεκτικά ε, συστήματα υγειονομικής περίθαλψης ε, που υπονοεί τη δυνατότητα πρόσβασης του πληθυσμού εκεί. Στο πλαίσιο αυτού τη ανακοίνωση ε, προσδιορίσαμε διάφορε διαστάσει τη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη όσον αφορά για το ποιο καλύπτεται, τι καλύπτεται, κατά πόσο οι τιμέ είναι προσιτέ, ε, αυτό σχετίζεται με τις συμμετοχές ε, που αναφέραμε προηγουμένως και ε, κατά πόσο είναι διαθέσιμη η φροντίδα όταν κάποιος βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση, υπάρχει διαθέσιμη υγειονομική περίθαλψη, υπάρχουν αρκετοί επαγγελματίε, ποιοι είναι οι χρόνοι αναμονής. Από αυτή την άποψη, η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη παρουσιάζει κενά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κενά που έγιναν ορατά κατά τη διάρκεια της κρίσης, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως εδώ. Δεν θα τα παρουσιάσω λοιπόν λεπτομερώς, αλλά ένα άλλο ζήτημα που παρουσιάζεται είναι ότι αν δει κανείς τους δείκτες, ακόμη και πριν την κρίση, ε, όπως και κατά τη διάρκεια της κρίσης, και εδώ κοιτάμε τους καλύτερους δείκτες που έχουμε στη διάθεσή μας όσον αφορά την πρόσβαση ε, στην υγειονομική περίθαλψη και είναι οι ανάγκες που δεν έχουν καλυφθεί. Το εξήγησε ήδη ο κύριος ε, Μπερτολίνη. Ε, τι σημαίνει αυτός ο δείκτης, οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες πηγαίνουν στους πολίτες και τους ρωτούν αν τους τελευταίους ορισμένους μήνες είχαν κάποια ανάγκη για κάποια εξέταση που δεν εκπληρώθηκε και ρωτάμε γιατί. Οι βασικοί λόγοι λοιπόν που δεν έχουν καλυφθεί αυτέ οι ανάγκε πρόσβαση στην οικονομική περίθαλψη είναι διαφορετικοί σε κάθε κράτο μέλο. Ε, και σε κάποια κράτη-μέλη υπάρχουν ζητήματα όσον αφορά τα δείγματα, για παράδειγμα, ή τι ερωτήσει τη έρευνα. Αλλά βλέπουμε παρόλα αυτά με μεγάλες ανισότητες μεταξύ συστημάτων. Ξέρετε, συνήθω ε, είναι πολύ δύσκολο να καλύψουν οι έρευνε τι ευάλωτε ε, ομάδε. Οπότε οι ανισότητε ενδέχεται να είναι χειρότερε από αυτέ που βλέπουμε εδώ σε αυτά τα γραφήματα. Στην επόμενη διαφάνεια, ε, την είδατε πριν δύο λεπτά, είναι, είναι πολύ σημαντική, όπω καταλαβαίνετε. Είχε συμπεριληφθεί στην γνωμοδότηση του πάνελ εμπειρογνωμόνων δεν ξέρω να γνωρίζετε αυτή την ε, γνωμοδότηση. Το 2013 η Επιτροπή ε, σύστησε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων για να διαρρευνήσει του αποτελεσματικού τρόπου επένδυση στην υγεία, αποτελούμενοι από ανεξάρτητου ε, εμπειρογνώμονε, στου οποίου ανήκει και ο κ. Λαμάτα, και πρόσφατα δημοσίευσε αυτό το πάνελ μια ε, γνωμοδότηση για την πρόσβαση στην υγειονομική περιθέλψη που ζήτησε η Κομισιόν και αυτό το γράφημα αποτελεί κομμάτι αυτή τη αρχική γνωμοδότηση. Η τελική γνωμοδότηση θα δημοσιευτεί σύντομα και σα παροτρύνω να τη διαβάσετε. Θα υπάρχει διαθέσιμη στο ιστοσελίδα του Πανέλ Εμπειρογνωμόνων όσον αφορά του αποτελεσματικού τρόπου πρόσβαση στην υγειονομική περιθέλψη και εκεί διαφαίνεται ότι οι ευάλωτε ομάδε επηρεάστηκαν ε, εντονότερα από την κρίση. Αυτό συμφωνεί φυσικά και με την κοινή λογική όσον αφορά τα οικονομίε μα και τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψη. Δείχνει και κάτι άλλο. Πολλά είναι τα προβλήματα όσον αφορά την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη. Ένα από αυτά είναι η δυσκολία καταμέτρησης, ε, ε, εκτίμησης ε, μαθηματικά του προβλήματο. Είναι πολύ δύσκολο να επιλεγούν οι δείκτε. Οι δείκτε που έχουμε δεν είναι πάντα συγκρίσιμοι και μετά υπάρχει άλλο ένα ζήτημα που αναφέρθηκε και προηγουμένω ότι τώρα δουλεύουμε με στοιχεία του 2013. Το πρόβλημα δηλαδή δεν είναι μόνο ε, ότι οι επιπτώσεις της κρίσης κάνουν χρόνο για να εμφανιστούν ε, στους δείκτες, αλλά ότι υπάρχουν και, υπάρχει και χάσμα μεταξύ ε, της παροχής ε, υπηρεσιών και των προβλήματων υγείας όταν συζητάμε για αλλαγέ του ΑΕΠ, για παράδειγμα, έχουμε στοιχεία του προηγούμενου, προηγούμενων ετών. Εδώ, στην προηγούμενη περίπτωση, είμαστε το 2016 και μιλάμε για τα δεδομένα ε, πρόσφατα στην υγειονομική υπεριθάλψη το 2013. Οπότε αυτό είναι ένα πρόβλημα. Για να σα εξηγήσουμε τι κάνουμε αυτή τη στιγμή όσον αφορά την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, το 2013 οι οργανισμοί ασθενών δραστηριοποιήθηκαν ε, έντονα όσον αφορά την πρόσβαση στην περίθαλψη και δημιούργησαν μία ε, έναν οργανισμό ε, εταιρικής σχέσης όσον αφορά ε, την πρόσβαση, όχι μόνο για τον ορισμό της πρόσβασης, αλλά και για την καταμέτρησή του, για την εκτίμησή του. Αυτό οδήγησε σε μια εταιρική σχέση που τώρα ε, αποτελεί πραγματικότητα και στην οποία συμμετέχουν πολύ ενδιαφερόμενοι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η DJ Health συμμετέχουν σε αυτές τις συζητήσεις. και αυτό οδήγησε στη δημιουργία μιας ομάδας ε, ενδιαφορμένων εδώ ε, μεταξύ βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, με θέμα την πρόσβαση στην περίθαλψη που απαριθμεί σήμερα περίπου 30 ευρωβουλευτές. Κάτι άλλο το οποίο μελετάμε και από το που έχουμε μεγάλες προσδοκίες είναι αυτή η γνωμοδότηση της ομάδας εμπειρογνωμόνων που θα είναι διαθεσμή σύντομα διότι διαπιστώσαμε ότι έχοντας δει ήδη την προκριτική γνωμοδότηση μπορεί να αποτελέσει πολύ καλή βάση για συζήτηση για να καθιερώσουμε ένα σωστό πλαίσιο ε, για τις συζητήσεις ε, πρόσβαση στην υγειονομική περιθέτωση και ταυτόχρονα συμβαίνουν διάφορα. Πέρυσι ε, στον προπολογισμό εγκρίθηκε ένα πιλωτικό έργο για την πρόσβαση στην υγειονομική περιθέψη σε αγροτικές περιοχές αυτό είναι ένα από του τομεί ε, όπου εντοπίζονται πολλέ ευάλωτε ε, ομάδε. Οι εργασίε έχουν ξεκινήσει. Μελετάμε και άλλα παρόμοια ε, παρεμφερή θέματα, προγράμματα. Παρεμπιπτόντω, το 2016 θα ξεκινήσει ένα άλλο πιλωτικό πρόγραμμα εκτίμηση τη πρόσβαση στο υγειονομική περιθαλψη. Είχε εγκριθεί στον προπολογισμό για το 2016 του Κοινοβουλίου. Οπότε από μένα γίνουν πολλές εργασίες ε, σε αυτόν τον τομέα. Τα αποτελέσματα είναι πρακτικής φύσης. Από το 2013, όταν ε, άρχισε να επιταχύνεται αυτή τη η εργασία, κάθε χρόνο βλέπουμε συστάσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου όσον αφορά την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, δηλαδή εκκλήσεις προ κράτη-μέλη να βελτιώσουν ή να συντηρήσουν την πρόσβαση ε, στην υγειονομική περίθαλψη ξεφεύγοντα από την καθαρά δημοσιονομική πτυχή τη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη όπω ε, συνέβαινε το 2012, όπου αναφερόμασταν μόνο σε αποτελεσματικό κόστο σε δημοσιονομικά ζητήματα. Από το 2013 λοιπόν, δηλαδή εδώ και τρία χρόνια, έχουμε συστάσει και για την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη. Ένα, μια άλλη ένδειξη είναι ότι αν δει κανεί ε, την ετήσια ε, έκθεση τη ανάπτυξη του 2016 που αποτελεί ένα έγγραφο πλαίσιο για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο ε, θα δείτε ότι εκεί αναφέρεται ρητά ότι η πρόσβαση στην υγειονομική περιθέλψη αποτελεί σημαντικό κομμάτι και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών οικονομιών. Ανισχύα που είχε εκφραστεί και εδώ. Νομίζω ότι αρχίζει να διαφαίνεται καθαρά ότι αποτελεί πλέον κομμάτι του θεματολογίου ως κομμάτι της βελτιωμένης ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής. Τώρα για το μέλλον όπως είπα, θεωρούμε ότι η βελτίωση της ε, ε, μέτρησης του υπολογισμού, της εκτίμησης της πρόσβασης ε, αποτελεί προϋπόθεση για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στον τομέα. Οπότε άμεσο στόχος μας είναι να, να βελτιώσουμε αυτή την εκτίμηση, να έχουμε συγκεκριμένους δείκτες, να βελτιώσουμε τους τρέχοντες δείκτες ή να βρούμε νέους Αλλά αυτό που είναι σίγουρο ότι χρειαζόμαστε δείκτε ε, κοινά αποδεκτού από όλου ενδιαφερομένου, ώστε να συζητάμε βάσει των ίδιων δεδομένων, να μπορούμε να εντοπίσουμε τα προβλήματα και να βρίσκουμε λύσει για αυτά. Φυσικά, στόχο είναι ε, πάντα να υποστηρίζουμε τα κράτη-μέλη ώστε να βελτιώσουν την πρόσβαση των πολιτών του σε καλή υγειονομική περίθαλψη με συνέπεια τη βελτίωση της υγείας των πολιτών μέσω της εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών ε, για ποιοτική υγειονομική περίθαλψη κάτι που θεωρούμε είναι πρωταρχική σημασία ε, για την ευρωπαϊκή κοινωνικο-οικονομική σύγκληση ως αποτέλεσμα των τελευταίων εξελίξεων ε, και όσον αφορά και των εκθέσεων ε, όπου διαφαίνεται αυτή η ιδέα πολύ καθαρά. Κάτι που έχει ήδη γίνει προς αυτή την κατεύθυνση είναι μια ομάδα εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση των επιδόσεων των συστημάτων υγείας όπου συμπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η Σουηδία. Σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την υποστήριξη και διεθνών οργανισμών όπως του ΠΟΕ, του ΟΣΑ και του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τις ε, πολιτικές υγείας. Ε, τα κράτη-μέλη μαζί με την Ορβηγία επίσης ε, συζητούν και συναντιόνται κάθε τρει μήνες για να συζητήσουν μεθοδολογίες και εργαλεία βελτίωσης των συστηματών υγείας τους. Όλοι ε, γνωρίζουμε ε, ότι οι συγκρίσεις και οι κατατάξεις το, συγκριτικά μεταξύ των συστημάτων των κρατών μελών είναι κάτι δύσκολο αλλά τα κράτη-μέλη συζητούν πώς μπορούν να εκτιμούν εσωτερικά τα ε, συστήματά τους και να συγκρίνουν μεθοδολογίες και εργαλεία. Πέραν αυτού, τα κράτη-μέλη έχουν συμφωνήσει κάθε χρόνο να υπάρχει ένα συγκεκριμένο θέμα προς συζήτηση. Το 2015 ήταν το έτος συζήτησης της ποιότητας και σύντομα θα δημοσιευτεί μια έκθεση για την ποιότητα της ε, ε, παροχής υγειονομικής περιθέλεψης από αυτή την ομάδα εμπειρογνωμόνων. Τώρα, η πρόσβαση στα φάρμακα είναι μία από τις διαστάσεις της πρόσβασης στην υγειονομική περιθέψη. Ουσιαστική γνωμοδότηση αυτής της ομάδας εμπειρογνωμόνων, αν τη διαβάσετε, θα δείτε ότι εντοπίζει οκτώ διαφορετικές διαστάσεις ε, της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και μια από αυτές είναι η πρόσβαση στα φάρμακα και στις ιατρικές συσκευέ. Έχω δύο διαφάνειες εδώ για να τελειώσω την παρουσίασή μου γιατί ευθυγραμμιζόταν με το θέμα του εργαστηρίου οπότε θεώρησα ότι θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και φυσικά σκοπός της Κομισιόν είναι να διασφαλίσει επιτυχή, ε, επιτυχή, επιτυχής θεραπείες σε προσιτές τιμές και να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις των ε, συστημάτων τιμολόγηση ε, με βελτίωση του συντονισμού και τις συνεργασίες, όπως είπαμε φυσικά ε, εδώ το έργο μας περιορίζεται λόγω των εθνικών αρμοδιοτήτων στο πλαίσιο της επικουρικότητας αλλά ε, αυτό που μπορεί να κάνει η καλύτερη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μπορεί να το πραγματοποιήσει με συνεργασία και συντονισμό με τα κράτη-μέλη. Γίνονται λοιπόν πολλά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτών. Πρώτα απ' όλα πρόσφατα χαρτογράφησε τις αρμοδιότητες στον τομέα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την πρόσβαση στα φάρμακα που προετοιμάστηκε από την ομάδα εμπειρογνωμάνων ε, για την δημόσια υγεία συγγνώμη, από την ομάδα εργασία ε, για την δημόσια υγεία είναι διαθέσιμο το έγγραφο αυτό στο Συμβούλιο και δείχνει την πολυπλοκότητα της διακυβέρνησης στα διάφορα κράτη-μέλη όσον αφορά την πρόσβαση στα φάρμακα. επίση μια ομάδα εμπειρογνωμόνων ε, επωνομαζόμενη ΣΤΑΜΠ για την ασφαλή και έγκαιρη πρόσβαση στα φάρμακα στην Κομισιόν συζητά ουσιαστικά το κομμάτι αυτό ε, μαζί με εμπειρογνώμονες ε, των ρυθμιστικών αρχών των κρατών μελών και εξετάζει τις αδειοδοτήσεις της ΕΜΑ και τις παρουσιάζει και τα συμπεράσματα στο Συμβούλιο. Μετά η Κομισιόν υποστηρίζει τα κράτη-μέλη μέσω μιας κοινής ε, δράσεις για την ε, αξιολόγηση της, των τεχνολογιών υγείας. Ε, κάτι που δημιουργήθηκε δύναμη της διατάξης βάση της οδηγίας 2011-2024 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. όλα αυτά φυσικά εξαρτώνται από τη βούληση συνεργασίας και συμμετοχής από τα κράτη-μέλη, αλλά υποστηρίζεται από την Κομισιόν. Επίσης έχουμε την απόφαση για τις δύο συνοριακές απειλές ε, που αφορά την κοινή προμήθεια ε, εμβολίων και άλλων ε, ιατρικών αντίμετρων. Είναι ένα ζήτημα το οποίο συζητείται τακτικά. Όπως είπα δεν χρειάζεται πάντα εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έχουμε δει παραδείγματα τεράστιων προμηθειών μεταξύ κρατών μελών και αυτό είναι καλό σημάδι. Μετά χρηματοδοτεί η Κομισιόν τη βελτίωση της Ευρωπαϊκής Βάσης Δεδομένων βάσει δεδομένων ε, τη οποία ε, συνεργάζονται τα κράτη-μέλη, γνωστοποιώντα το ένα στο άλλο τι τιμέ των φαρμάκων. Και η μεγαλύτερη αναγκαίκη είναι βελτίωση του σημερινού συστήματο. Ε, θα βοηθήσει μάλλον αυτή η βάση δεδομένων να βελτιωθεί, ε, να βελτιωθεί η λειτουργία των σημερινών συστημάτων. Ε, πολλά κράτη-μέλη συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα, καθώς και άλλοι ενδιαφορόμενοι οι τομείς, ε, τις ε, οργανώσεις ασθενών και ευρωβουλευτές συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα και τέλος αυτή τη στιγμή διεξάγουμε μια μελέτη για βελτιωμένο συντονισμό μεταξύ χωρών για την τιμολόγηση βασίζεται σε μια μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2004 θέλουμε να βελτιώσουμε την ανάλυση που γίνεται σε αυτή τη μελέτη και να εξετάσουμε πιθανούς ε, μηχανισμούς ε, όπως ε, διαφοροποίηση της τιμολόγησης και συντονισμό. Βρίσκεται σε φάση τελικού σχεδίου, λογικά θα λάβει την οριστική της μορφή σε μερικούς μήνες. Κάνα δύο μήνες μάλλον. Αυτά είχα να σας παρουσιάσω σήμερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Να δώσουμε τώρα το λόγο στους συναδέλφους. Πρώτος ο συνάδελφος ε, Κόφολη. Ε, ευχαριστώ. Επανελήφθη η έννοια ότι το θέμα είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρω είναι. Βέβαια, ε, αυξάνεται το κόστος. Έχουμε τη γύρανση της Ευρώπης. Γερνά η Ευρώπη κοστίζουν οι νέες τεχνολογίες. Ε, αληθεύει ότι αυτή η κρίση οδήγησε σε αύξηση των διαφορών και των ανισοτήτων εντός των χωρών και μεταξύ χωρών. Αυτό είναι το θέμα. Βλέπουμε και σήμερα στην περίπτωση των φαρμάκων σπατάλες και καταχρήσεις. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να εργαζόμεθα όπως κάνουμε, να προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε την κατάχρηση του αλκοόλ, του καπνού και να κάνουμε και εκστρατείες και προσπάθειες κατά των δαπανών, των σπαταλών και των ε, καταχρήσεων των φαρμάκων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θα πρέπει να ευνοήσουμε τις επενδύσεις για την πρόληψη και την παιδεία. Και η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία. Και αυτό πιστεύω ότι είναι ένα πεδίο δράσεως ε, που πρέπει να κάνουμε κάτι στον τομέα σαν Ευρωπαίοι. Σήμερα μιλάμε για κυκλική οικονομία. Θέλουμε να κάνουμε περισσότερα με λιγότερα. Θέλουμε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης. Και στον τομέα αυτό της πατάλης στα φάρμακα, όλα τα φάρμακα που δεν έχουν λήξει και πετάγονται Έχουμε αύξηση ε, και σε αυτά αποβλήτως σε αυτό τον τομέα. Ε, υπάρχει σπατάλη. Λοιπόν, και αυτό μπορούμε να το σκεφτούμε και να το εξετάσουμε. Χρειάζεται μια ευάθυνση και αυτό το κομμάτι. Κατά την άποψή μου υπάρχουν περιθώρια σημαντικά οικονομιών εκεί. Ευχαριστώ κύριε Κόφολη. Η κυρία Κίρτον Ντάρλινγκ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ για τους τρεις ομιλητές μας. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση όλη η έρευνα που γίνεται για την καινοτομία στον φαρμακευτικό κλάδο και ότι πολλοί από την έρευνα και ανάπτυξη γίνεται απευθείας από τις φαρμακευτικές ενώ ορισμένοι οικονομολόγοι όπως η Μαρία Ματσουκάτου λένε ότι κυρίως το κράτος κάνει την περισσότερη καινοτόμα έρευνα στο φαρμακευτικό τομέα και απλώς οι φαρμακευτικές εταιρείες ε, κάνουν μικροαλλαγές στα φάρμακά τους για να διατηρηθεί η αποκλειστικότητα και άρα τα κέρδη τους. Δεν ξέρω αν το βλέπετε από διαφορετική οπτική γωνία. Θα ήταν ενδιαφέρον όμως να δούμε πώς αυτή η συζήτηση επηρεάζει τη δημόσια πολιτική για την υγεία και για την ε, τιμολόγηση. Θεωρώ ότι το σημαντικότερο είναι η διαφάνεια για να μην υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόντων, να μην υπάρχουν εγκατεστημένα συμφέροντα που επηρεάζουν το καθορισμό των τιμών. Είμαι στην Ίντα και αυτό είναι ιδιαίτερα επίμαχο. Για παράδειγμα στην διατλαντική εταιρική σχέση Γίνεται μεγάλη συζήτηση εκεί για την τιμή των φαρμάκων. και για τις σχέσεις μας με τις χώρες της Βόρειας Αμερικής. Υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία, έγινε μια προσπάθεια να ενημερωθεί η οδηγία για τη διαφάνεια του 89, αλλά δυστυχώς δεν έχει περάσει το Συμβουλίο. Και από ό,τι καταλαβαίνω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την έχει αποσύρει εντελώς τα πλαίσια του θεματολογίου για καλύτερες ρυθμιστικές διατάξεις. Θέλετε περισσότερη πίεση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε αυτή την νομοθεσία για να διασφαλίσουμε την διαφάνεια. Η Σολεδά είχε υποβάλει μια προφορική ερώτηση πέρυσι τον Ιανουάριο στην Επιτροπή. Ρωτούσε τι μέτρα θα ληφθούν ούτως ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια. Και η απάντηση της ε, Επιτροπής ήταν ότι κάτι ετοιμάζουμε. Ε, θεωρώ ότι αυτά που είπε ο κύριος Καρβάλιο για ένα task force και μια κοινή προσπάθεια και τη μελέτη που είναι σε φάση εκπόνησης ότι εντάσσεται στην ίδια προσπάθεια αλλά θεωρείται ότι στην πράξη έχει υπάρξει καμία επίπτωση. Υπάρχει καλύτερη, για παράδειγμα, ενημέρωση μεταξύ κρατών μελών για τις τιμές των φαρμάκων. Υπάρχει κάτι θετικό. Και κάτι άλλο για το οποίο ήθελα την άποψή σα. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε τη χρήση των γενοσύμων στην Ευρώπη. Ορίζον 2020 μπορεί να βοηθήσει για τις συνθήκε έρευνας και ανάπτυξης όταν συμμετέχει ο δημόσιος τομέας στην φαρμακευτική έρευνα και κάτι ακόμη. Τι ρόλο μπορούν να παίξουν ε, οι κοινέ αγορές, οι κοινέ προμήθειες φαρμάκων. Ότι είδαμε για παράδειγμα ότι η Ολλανδία και το Βέλγιο αγοράζουν από κοινού φάρμακα για να επιτύχουν καλύτερες τιμές. Ε, θα μπορούσαμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να κάνουμε μια προσπάθεια για κοινέ προμήθειες. Ευχαριστώ. Μπεθέρα. Αλλά παρακαλώ συντομία για να έχουμε χρόνο να ακούσουμε και τις απαντήσεις γιατί 12.30 ε, πρέπει να φύγουν οι διερμηνείς. Καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω τους εισηγητές. Μα τι σημαίνει. Ευχαριστώ τον κύριο Λαμάτα για τις συγκεκριμένες προτάσεις του νομίζω ότι έκανε μια σαφέστατη ανάλυση και πολύ συγκεκριμένη πρόταση που πλήρως υποστηρίζω. Είναι απαράδεκτες οι μονοπωλιακέ καταστάσεις για λόγους αποτελεσματικότητα πάνω απ' όλα. Δεν λειτουργεί. Δεν εξυπηρετεί τον στόχο για τον οποίο δημιουργήθηκε. Πρέπει να αλλάξει. Αν δεν εποφελείται η κοινωνία από κάτι πρέπει να αλλάζει. Και όχι μόνο έχει απαράδεκτε παρενέργειε για την πρόσβαση στην υγεία, αλλά εξυπηρετεί άλλους σκοπούς. Αυτή η πρόταση για μια κοινή ευρωπαϊκή πλατφόρμα είναι εφικτή και πολύ καλή. Μέσω των αντιβιωτικών. Νομίζω ότι είναι σκόπιμο να αρχίσουμε. Να αρχίσουν από εκεί τα εργαστήρια γιατί τα αντιβιωτικά δεν είναι πάνω-πάνω από πλευρά τιμών. Και γιατί τα αντιβιωτικά και η αντίσταση στα αντιβιωτικά είναι σοβαρό πρόβλημα δημόσια υγεία. Συμφωνώ λοιπόν πλήρω Θα ήθελα να μπορέσουμε να παίξουμε ρόλο εμείς για να ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια. Ευχαριστώ τον κύριο Μπερτολίνη που τόνισε ότι η υγεία είναι πολιτική επιλογή και τις επιλογές τις κάνουμε εμείς. Και ανάλογα με τις επιλογές είναι και τα αποτελέσματα. Και βεβαίως πρέπει να παίξουν ρόλο όχι μόνο οι εθνικές κυβερνήσεις με την επικουρικότητα που όλοι αναγνωρίζουμε, αλλά και η Ευρώπη θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Καρβάλιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί ξέρετε η παρουσίασή του θα μπορούσε να δώσει την εντύπωση ότι, ότι η Κομισιόν τα λέει μεταξύ της. Δεν έχει καμία δυνατότητα να επιδράσει ως πολιτικό όργανο διαχείρισης της Ένωσης εντός των περιορισμών που τίθενται στην ε, λειτουργία της. Έχει δυνατότητα η Κομισιόν να ε, προκαλέσει αποφάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν αυτή την αλλαγή προτύπου. Για παράδειγμα, αποφάσεις που αφορούν τη χρηματοδότηση και τι ε, επιστροφή, τι, τι κέρδος περιμένουμε να προκύψει από αυτά τα καινοτόμα ε, φάρμακα και το κέρδος πρέπει να είναι και καλύτερη πρόσβαση και για τους πολίτες ή μέσω κοινών προμηθειών ή μέσω της ε, παραγωγής ε, και ε, χορήγησης γενοσύμων όταν υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας. Όπως είναι η μεσω της παραγωγης και χορηγησης γενοσυμων οταν υπαρχει ενα σοβαρο προβλημα δημοσιας υγειας οπως ειναι η πατητη C που θεωρούμε ότι μπορεί να αφορά 9 εκατομμύρια ασθενείς. Πρέπει λοιπόν να υπάρξουν συγκεκριμένες ενέργειες και η Κομισιόν κατά τη γνώμη μου πρέπει να παίξει ηγετικό ρόλο. Και εμείς ως Κοινοβούλιο ήδη το προσπαθούμε και θα συνεχίσουμε να το επιχειρούμε. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφε Πεθάρα. Η συνάδελφος ήδη σύντομα παρακαλώ πολύ γρήγορα περισσότερο σκέψη και να εκφράσω κάποια ανησυχία ακούγοντα αυτό το τελευταίο κομμάτι του πάνελ. Οι ομιλίε που έξω ήταν οι παρουσιάσει ήταν πολύ ενδιαφέρουσε, αλλά μου δημιουργούν ανησυχίε. Διαφαίνεται ότι ε, κατά καιρούς ε, το κέρδος ε, υπερισχύει του συμφέροντος των πολιτών. Χρησιμοποιούμε εργαλεία αγοράς για να επιλύσουμε πάντως τους προβλήματα του περιβάλλοντος, της υγείας, όλες τις τύχες ζωής μας και μου έρχεται στο νόμο η Ιταλία όπου μόλις 250 υπηρεσίες δόθηκαν από τη Δημοσιαρχή Υγείας και ιδιωτικοποιήθηκαν. Δηλαδή μιλάμε τώρα ε, τι μέτρα πρέπει να λάβουμε για να προστατεύσουμε την υγεία των πολιτών και να αποφύγουμε να ευνοείται η άνθηση λύσεων ε, του ιδιωτικού τομέα. Αυτή είναι μια σκέψη που θέλω να σας θέσω. Βλέπετε ενδείξεις πραγματικά θετικές ή μήπως ε, εξακολουθούμε να παίζουμε το ίδιο παιχνίδι χωρίς να λύνουμε ποτέ κανένα πρόβλημα και χωρίς να τα ποτέ. Ένα λεπτό, Ένα λεπτό, Πέντερ, παρακαλώ. Δεν θα παραλάβω αυτό που υπόθηκαν δύο προτάσει για εμά τους ίδιου. Πρώτον, η Επιτροπή Έρευνας, συγγνώμη, η Επιτροπή Αναφορών, πρέπει να απαιτεί κοινωνική ρήτρα πάντα σε όλα όσα κάνει. Όλοι πρέπει να έχουν πρόσβαση στο σύστημα υγεία. Αυτό να το λάβουμε υπόψη στι απαντήσει στι αναφορές και να βλέπουμε εάν τηρείται αυτή η κοινωνική ρήτρα. Και επίση πρέπει να κάνουμε πολλά κι εμεί και η γραμματεία αυτές προτάσεις που έγιναν και οποιαδήποτε θετική δυνατότητα να τις ε, στείλουμε στις ε, αρμόδιες επιτροπές. Είναι πολύ σημαντικό γιατί δεν θα πρέπει να λήξει με τη σημερινή ακρόαση η συζήτηση, θα πρέπει να είναι σημείο αφετηρίας. Πρέπει να υπάρξουν και νομοθετικές πρωτοβουλίες με τις οποίες να ασχοληθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ Πέτερ. Να δώσω τώρα το λόγο στους ομιλητές μας. Και αν υπάρχει δυνατότητα θα κάνω και εγώ κάποιες καταληκτικές παρατηρήσεις. Αλλά πρώτα λοιπόν εδώ στους ομιλητές μας. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο κύριος Λαμάτα. Να ξεκινήσουμε την τελευταία παρατήρηση. Είναι βεβαίως Αυτή η ζήτηση πρέπει να έχει συνέχεια. Υπόθηκαν συγκεκριμένα πράγματα ε, εδώ στα γρήγορα. Αλλά το θέμα αυτό ε, ενδιαφέρει πολύ τους ε, πολίτες. Έχουν κάνει αναφορές που θέλουν να λάβουν απάντηση. Άρα πρέπει να δοθεί απάντηση ανάλογα με τις αρμοδιότητες των ΜΕΝ και των ΔΕ. Ε, ορισμένοι εξέφρασαν κάποια απεσιοδοξία. Αντίθετα, πρέπει να την μετατρέψουμε σε κάτι θετικό. Το σύστημα υγείας, το δημόσιο σύστημα υγείας έχει βελτιωθεί καθ' όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα και είναι υπόδειγμα. Το κοιτάνε με θαυμασμό στον κόσμο, αλλά έχει προβλήματα, υφίσταται απειλές αλλά ε, το θέμα είναι πώς θα τα επιλύσουμε αυτά, πώς θα εξακολουθήσουμε να βελτιώνουμε την κατάστασή του. Για το μέλλον, συμφωνώ με αυτά που μόλις υπόθηκαν, το μέλλον είναι δημόσια υγεία, είναι η πρόληψη, είναι να υπάρξει περισσότερη αποτελεσματικότητα στα πλαίσια των υφισταμένων πόρων. Αυτή είναι η μεγάλη προσπάθεια του 21ου αιώνα. Η Ευρωπαϊκή, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρμοδιότητα, όπως ήδη υπόθηκε, μπορούμε να αξιοποιήσουμε το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο εντός του οποίου έγιναν πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Υπήρξαν συγκεκριμένες συστάσεις για τα συστήματα υγείας, για να βελτιωθεί για παράδειγμα η πρόσβαση ή η διαχείριση της προμήθειας φαρμάκων. Η Ευρώπη λοιπόν αξιοποιεί την κρίση ως ευκαιρία για να βελτιώσει την κατάσταση μέσω εξέτασης του τι έχει γίνει και οι ετήσιες εκθέσεις ε, ανάπτυξης μπορούν να μας βοηθήσουν. Για την έρευνα, βεβαίω, 50% της έρευνας ήδη χρηματοδοτείται δημοσίως μέσω πανεπιστημίων, ε, ε, επιδοτήσεων κτλ. Και το υπόλοιπο είναι ιδιωτικό. Αυτό πρέπει να συζητήσουμε. Όπως είπε και η Μαριάννα Ματσουκάτσου, στις περισσότερες περιπτώσεις τα καινοτόμα φάρμακα προέκυψαν μέσω άμεσης δημόσιας χρηματοδότησης. Πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε να το εξετάζουμε αυτό και γι' αυτό το θέμα έχει αρμοδιότητα ένωση γιατί χρηματοδοτεί προγράμματα έρευνας που θα μπορούσε να ε, απαιτήσει να είναι πιο αποτελεσματικά μέσω μιας ε, δημόσιας πλατφόρμας έρευνας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την ε, συζήτηση. Ε, Τέτοιαν πολύ σημαντικά θέματα. Δύο σχόλια πρώτα απ' όλα όσον αφορά την ε, κατάχρηση των φαρμάκων και τη σπατάλη που ανέφερε ο κ. Τζόφολη στην αρχή και την έμφαση στην πρόληψη. Φυσικά είναι πολύ σημαντικό ζήτημα και έχει επιπτώσεις και για το κόστο, αλλά είναι και σημαντικό ζήτημα και για την αντιμικροβιακή αντίσταση που αποτελεί όλο και μεγαλύτερο ζήτημα για την Ευρώπη αλλά και εκτός. Η αντιμετώπιση λοιπόν τη σωστή ε, χρήση των ε, φαρμάκων και η αποφυγή αυτού του είδου των προβλημάτων, των προβλημάτων αυτού του είδου θα βοηθήσει να ε, αντιμετωπίσουμε και το ζήτημα τη μικροβιακή αντίσταση που είναι κρίσιμη σημασία. Εδώ αυτή η πρόταση δημιουργίας μιας ερευνητική πλατφόρμας, εντάξει τώρα δεν μιλώ επίσημα, βέβαια το λέω προσωπικά, είναι καλή πρόταση κατά την προσωπική μου άποψη γιατί πρέπει να ενθαρρύνουμε ε, δημόσιες και ιδιωτικές πρωτοβουλίες για την πρόθεση και την εξέβριση νέων φαρμάκων, ειδικότερα στον τομέα των αντιβιωτικών που αρχίζει να αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία ανησυχίας μας για τα επόμενα χρόνια. Ένα μικρό σχολείο για την αισιοδοξία, την απεσιοδοξία. Ε, Συμφωνώ με το όσο είπε ο καθηγητή ο κ. Λαμάτα προηγουμένω. Η υγεία έχει σημειώσει τεράστιε πρόοδου στι τελευταίε δεκαετίε στην Ευρώπη και αυτό είναι σημαντικό. Πρέπει να υποθεί. Αλλά πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα ζητήματα υγεία και τα κοινωνικά ζητήματα θα είναι κομμάτια τη συζήτηση ε, όταν οι κυβερνήσει λαμβάνουν σημαντικέ αποφάσει οικονομική ανάπτυξη. Πιστεύω ότι ε, τι τελευταίε δεκαετίε η συζήτηση στην Ευρώπη έχει περιοριστεί ε, σε μακροοικονομικά θέματα χωρίς να λαμβάνονται υπόψη όλες αυτές οι παρενέργειες ε, ορισμένων επιλογών. Πιστεύω μια σοφή προσέγγιση ε, για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος και ένας διάλογος με τον οικονομικό τομέα θα βοηθήσουν να ληφθούν όλα αυτά υπόψη. Διότι αυτή τη στιγμή εγώ παρακολουθώ τη συζήτηση σε διάφορες χώρες και στη δική μου ειδικότερα αλλά δεν βλέπω να λέγεται και τίποτα για να αποτελούν κομμάτι των συζητήσεων ή των διαδικασιών λήψη αποφάσεων ε, τέτοια θέματα. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό και εκτιμώ ιδιαίτερα αυτή τη συζήτηση που κάναμε εδώ στην Επιτροπή Αναφορών. Είναι μια από τις πρώτες φορές που βλέπω να ε, βλέπουμε ε, υπό αυτό το πρίσμα το πρόβλημα αυτό. Ελπίζω να συνεχιστούν αυτές οι συζητήσεις και στο μέλλον. Thank you. Um, on the capacity of the... Ευχαριστώ. Όσον αφορά την ικανότητα της Κομισιόν να κάνει περισσότερα ε, για θέματα υγείας, πιστεύω ότι οι συνθήκες ε, καθορίζουν επακριβώς τις εθνικές αρμοδιότητες για την υγεία. Και αυτό φυσικά θέτει περιορισμού ε, στι αρμοδιότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δίνει και στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να μπλοκάρουν πράγματα που έχουν ολοκληρωθεί. Θα μπορούσαν να γίνουν εύκολα. Παρ' όλα αυτά έχει κάνει πολλά για την υγεία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, για παράδειγμα, είναι πολύ σημαντικό σήμερα. Οι ευρωβουλευτέ μίλησαν επίση για, για την πρωτοβουλία καινοτόμων φαρμάκων. Να αναφέρω επίση ε, και την οδηγία για τα δικαιώματα ε, σε θέματα διασυνοριακή ε, υγειονομική περίθαλψη ή για την κοινή δράση για τι τεχνολογίε υγεία. Είναι ουσιαστικά δύο πρωτοβουλίε που βρίσκονται σε πρώιμα στάδια αλλά χρειάζονται την υποστήριξη των κρατομένων για να επιτύχουν. Συνεπώ αυτό αποτελεί σταθερά ένα περιορισμό για εμάς, αυτοί οι περιορισμοί που ε, θεσπίζει, θεσπίζουν οι συνθήκε. Και συμφωνώ με τον κύριο Λαμάτα για την σπουδαιότητα του Ευρωπαϊκού Εξωμήνου και ότι πρέπει να επισημάνουμε ότι η πρόσβαση και η ποιότητα τη ε, υγειονομική περίθαλψη πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με στα επόμενα χρόνια, ό,τι και να γίνεται. Ε, τώρα, όσον αφορά τι ερωτήσει που αφορούν την ανταλλαγή πληροφοριών ε, για, την, για τι τιμέ, για την τιμολόγηση και τι μπορεί να γίνει για να βελτιωθεί, τώρα από καθαρά άποψη οικονομική ανάλυση, το σημερινό σύστημα, το οποίο όπω εξηγήθηκε βασίζεται σε μονοπόλια, ε, νομικά μονοπόλια που δεν θα συζητήσω κατά πόσο είναι καλά ή κακά. Έχει ήδη συζητηθεί εδώ. Αλλά πιστεύω ότι η ανταλλαγή πληροφοριών είναι ο καλύτερο τρόπο για να βελτιώσουμε το τρέχον σύστημα, διότι το σύστημα αυτό χαρακτηρίζεται από ασυμμετρία πληροφοριών. Δηλαδή, το τομέα παραγωγή διαθέτει όλε τι διαθέσιμε πληροφορίε και αν τα κράτη-μέλη δεν μοιράζονται μεταξύ του τι πληροφορίε, όχι μόνο οι προφορές αυτές αποτελούν, ε, βρίσκονται στην κατοχή μόνο των ε, βιομηχανιών παραγωγής, αλλά και τα κράτη-μέλη έχουν μόνο τις δικές πληροφορίες και μερικές φορές και εντός του ίδιου κράτους μέλους ε, έχουμε... δεν γίνεται ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ περιοχών συγκεκριμένων νοσοκομείων. Δηλαδή υπάρχει μια ασυμμετρία δυνάμεων λόγω της ασυμμετρίας των πληροφοριών. Το πρόγραμμα για το οποίο σα εξήγησα αποτελεί μια ανταλλαγή πληροφοριών με τη συμμετοχή 26 κρατών μελών, αλλά εδώ μιλάμε για ανταλλαγή πληροφοριών επί επίσημων τιμών. Αλλά ξέρετε τώρα επιμέρου, περιοχέ, επιμέρου νοσοκομεία μπορεί να επιβάλλουν άλλε τιμέ. Και αυτέ οι πληροφορίε δεν, δεν υπάρχουν στη διάθεσή μα. Όταν λοιπόν ένα κράτο μέλο ή ένα νοσοκομείο δια... κάνει διαπραγματεύσει, δεν γνωρίζει ποιε είναι οι τιμέ σε άλλα νοσοκομεία, σε άλλε περιφέρειε, σε άλλα κράτη-μέλη όπου η βιομηχανία επειδή έχει μονοπόλιο σε μια συγκεκριμένη αγορά ε, τη συγκεκριμένη εποχή ε, έχει στη διάθεσή τη όλε τι πληροφορίε. Αν θέλουμε λοιπόν να βελτιώσουμε το σημερινό σύστημα, αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών. Εάν δούμε αν θέλουμε κάποιο άλλο σύστημα. Αυτό είναι κάτι πολύ ευρύτερο από την υγεία. Ακόμη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπω φαντάζεστε, θα έχει επιπτώσει στα δικαιώματα διανοητική ιδιοκτησία, στο εμπόριο, στο ανταγωνισμό στι πολιτικέ εσωτερικέ αγορέ. Είναι μεγάλη λοιπόν η συζήτηση. Δεν είναι κάτι που αφορά μόνο την υγεία. Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή του να αλλάξουμε το σημερινό σύστημα. Ευχαριστώ. Και εγώ σα ευχαριστώ όλου για να καταλήξω. Ευχαριστώ και πάλι τους ψυχητές Και τονίζω ότι θέσαμε όλοι το θέμα διαχωρισμού αρμοδιοτήτων. Γιατί ορισμένοι λένε έχουμε τη δυνατότητα, έχουμε τις δυνατότητες, έχουμε τα μέσα για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις. Εγώ νομίζω ότι Μπορεί να μην έχουμε με την αυστηρή έννοια την αρμοδιότητα, γιατί τα εθνικά συστήματα υγείας είναι εθνικά, αλλά έχουμε υποχρεώσεις δημόσιας υγείας ή μπορούμε να μιλήσουμε για τα θέματα αδειοδότησης για τα, φάρμακα, τα Διότι αυτά τα θέματα θίγονται και επηρεάζονται από πολλά, από πολλούς άλλους τομείς, οικονομικούς και μη. Άρα εμείς ως πολιτικοί πρέπει να επιβάλλουμε τις βασικές αρχές της καθολικότητας, της αλληλεγγύης, της ισότητας και πρέπει να πάρουμε τα αναγκαία μέτρα για να ανταποκριθούμε σε αυτές τις προκλήσεις. Συμφωνώ μαζί σας ότι ήταν σύντομη αυτή η συζήτηση, αλλά ήταν επί της ουσίας. Και το βασικό είναι να στείλουμε τα σωστά μηνύματα. Όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε σοβαρέ προκλήσει, ε, βέβαια είναι μόνο μια αφετηρία, θα συνεχίσουμε το διάλογο. Αλλά αποκομίζω μια πολύ καλή εντύπωση Καταλήξαμε σε σκόπιμα συμπεράσματα, ακούσαμε επίσης τον εκπρόσωπο της Κομισιόν και με χαροποίησε. Γιατί όσοι εργάζονται στις, ε, στους ευρωπαϊκούς θεσμούς ξέρουμε ότι τα πράγματα δεν προχωρούν όσο γρήγορα θα θέλαμε. Ξέρουμε ότι αυτό είναι αναγκαία επίπτωση της πολυμορφίας μας και του αριθμού των κρατών μελών που απαρτίζουν την Ένωσή μας. Είναι φυσιολογική αυτή η βραδίτητα αλλά με χαροποιεί ότι εργάζεται για το θέμα αυτό η Κομισιόν, άρα η ομάδα εργασία μας, εργασίας μας, όπως και παρόμοιες που είχαμε στις προηγούμενες θητείες, ευαισθητοποιούν για τα θέματα αυτά και βοηθούν να ληφθούν οι αποφάσεις. Οπότε εγώ θα φύγω από αυτή την ε, εκδήλωση με πολύ θετικές εντυπώσεις και θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανό ότι βήμα το βήμα θα καταλήξουμε στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Ευχαριστώ τους διοργανωτές. Σας ευχαριστώ όλους. Η εργασία που έγινε είναι πολύ σημαντική, δεν πήραν όλοι το λόγο, αλλά επίσης ε, η Μαρτίνα μας βοήθησε πάρα πολύ. Ευχαριστώ για τη δέσμευσή σου, την προσπάθεια, τις προσπάθειές σου, τις επαφές που έκανες. Σας ευχαριστώ όλους για την θαυμάσια εργασία που κατέστησε να χάρη, χάρη σε όλους σας. Ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά όλους.